Dear colleagues, good afternoon. you want to take your seats. Παρακαλώ συνάδελφοι καθίστε. This is being a long ongoing session of the Libe Committee. We got started. Ξεκίνησαμε χθες το πρωί στις 9 και σήμερα το απόγευμα είναι η τέταρτη σύνοδος της Επιτροπής μας μεικτή συνεδρίαση, ΛΥΜΠΕ και Επιτροπή Γυναικών. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Καλωσορίζω τον πρόεδρο της Επιτροπής ΦΑΜ, τον κύριο Γκούσταυσον, που βρίσκεται εδώ για να εξετάσουμε το σημείο 16 της Μεζίδης Διατάξεως που αφορά τους ελάχιστους κανόνες αναφορικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας. Έχουμε δύο συγητές από πλευράς ΛΥΜΠΕ, κυρία Τερέζα Χιμένας ε, Μπεσερίλ Μπάριο και από την ΦΑΜ η κυρία Αντωνία Παρβάνοβα. Έχουμε να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Σύγχρονα το, το έγγραφα και θα ορίσουμε και την προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών για να περάσουμε σε αυτό το δύσκολο έργο το οποίο μέχρι τώρα έχει αποδώσει ο κύριος Γκούσταυσον, ε, πρόεδρος της Επιτροπής ε, Γυναικών, θα λάβει το λόγο. Θα μιλήσω σου ειδικά. Ε, precis ε, Uh, uh, Ακριβώ όπω είπε ο πρόεδρο Ακυλάρ, έχουμε πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στι δύο επιτροπέ μα και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτό. Έτσι καταφέρνουν να καταλήξουμε σε αποτελέσματα όπω αυτό βλέπετε μπροστά σα. Στην πρόταση αυτή μπορεί να πει κανεί ότι υπάρχουν πολλέ πρόσθετε προτάσει, αλλά ε, θα πρέπει να το θεωρήσουμε αυτό δείγμα του πολύ μεγάλου ενδιαφέροντο που υπάρχει δεν σημαίνει ότι δεν είναι καλή η πρόταση που έχουν υποβάλει οι συγητέ. Είναι πάρα πολύ καλή δουλειά που έχουν κάνει οι συγγητέ. είναι εξαιρετική. Ε, το ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες, πολλές ε, προτάσεις για προσθήκε, δείχνουν το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το ενδιαφέρον αυτό. Η ύπαρξη πολλών τροπολογιών ε, ενισχύει το θέμα αυτό και έχω προσθήσει ότι υπάρχουν πάρα πολλέ προτάσεως για προσθήκες που ε, τονίζουν τα ε, μέτρα κατά της ε, βίας εξαιτίας του φύλου. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε καλή συνεργασία και την επόμενη εβδομάδα να ψηφίσουμε αυτήν την πολύ σημαντική ε, έκθεση. Ξαναδίνω το λόγο στον Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Κούσταυσον. Ναι, πράγματι. Έχουμε συνεργαστεί επανειλημμένα και το ξανακάνουμε τώρα. Αφού ακούσουμε τους εισηγητές, θα δώσουμε το λόγο στα άλλα θεσμικά όργανα, την ε, Επιτροπή και, και το Συμβούλιο και θα θέσουμε και η ημερομηνία για την ψηφοφορία. Θα συζητήσουμε το θέμα αυτό. Ας αρχίσουμε πρώτα την ε, κυρία Χιμένες Πεθερίλ που είναι η πρώτη ε, εισηγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Sí, eh, yo dejaría hablar primero a la señora Μήπως ε, να λάβει το λόγο πρώτα η κυρία Παρμανόβα, διότι στην προηγούμενη συνεδρίασή μας ε, έλαβα εγώ πρώτη το λόγο. Για λόγους αυρότητας λοιπόν, καταλαβαίνετε, θα προτιμούσα να λάβει το λόγο πρώτα η συνάδελφος. Ευχαριστώ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Κυρία Παρμανόβα έχει το λόγο. Uh, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Χιμένεθ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε για αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο και πολύπλοκο θέμα, αλλά να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους, τους και όλους τους συγκητές, όλους ιδιαίτερους, για τις 500 τροπολογίες που λάβαμε. Οι περισσότερες τροπολογίες ε, ευθυγραμμίζονται με τη βασική φιλοσοφία που θέλουμε να διέπει την έκθεση να ευχαριστήσω την Άντζελα, τη Ρομπέρτα από τη Γραμματεία της Επιτροπής Γυναικών, οι οποίες προσπαθούν από κοινού μαζί μας να καταλήξουν σε συμβιβαστικές τροπολογίες για να διευκολύνουν τη ζωή των μελών και των διεπιτροπών και να φτιάξουν ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλογο ψηφοφορίας που θα αρέσει σε όλους. Θα ήθελα να εστιάσω την προσοχή σας στα βασικά σημεία τα οποία θεωρούμε σημαντικά σε αυτή την έκθεση και επί των οποίων επικεντρώνεται και περισσότερε τροπολογίε. Πρώτα απ' όλα, ορισμοί. Ο βασικό στόχο ήταν ε, να έχουμε ένα συνεκτικό ορισμό που θα εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. κοινού με την κυρία Χιμένεθ και τα μέλη τη Επιτροπή ε, ΦΕΜ. Προσπαθήσαμε να λάβουμε υπόψη μας ε, τη δυναμική ε, του φύλου στα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικότητα και έχουμε δύο ορισμού. Ο πρώτος αφορά ε, την τη βία λόγω φύλου και την βία σε στενές σχέσεις. το έχει τόσο το θύμα, αλλά το δράστη και του έδωσε του εγκλήματος. Τονίσαμε επίσης και την ε, βία κατά των γυναικών. Λαμβάνοντα υπόψη και τη Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την πρόληψη και καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών. Η οδηγία είναι ένα οριζόντιο εργαλείο. Πιστεύουμε ότι ο πρώτο ορισμό ε, για τη βία ε, που βασίζεται στο φύλλο θα πρέπει να είναι ο ορισμός σε ό,τι αφορά το φύλλο, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να δίνει έμφαση στο δυσανάλογο αντίκτυπο τη βία πάνω στι γυναίκε. Γι' αυτό ρητά στον ορισμό αναφέρουμε ότι επηρεάζει ένα άτομο λόγο της ταυτότητας του φίλου και της έκφρασης του φίλου, αλλά δυσανάλογα πιο πολύ ε, θίγει τις γυναίκες. Η βίστορα τώρα για τη βία στις στενές σχέσεις. Εκεί δίνουμε έμφαση στη σημασία και της οικονομικής εξάρτησης. τη κοινωνική καταπίεση και άλλων οφών καταπίεση τη γυναίκα. Κάτι άλλο το οποίο συζητήσαμε ήδη είναι τα θύματα με ιδιαίτερε ανάγκε, με ειδικέ ανάγκε. Εμεί αναπτύσσουμε εδώ την ιδέα σε στενή συνεργασία και με τι ατομικές, μάλλον σε και με αξιολογήσεις, δηλαδή αντί να καταρτίζουμε κριτήρια ή να έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ στην οδηγία αυτή, θέλουμε να δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αναπτύξουν τα δικά του κριτήρια, αλλά πάντοτε δίνοντα προσοχή στα θύματα που ενδέχεται να απαιτούν ιδιαίτερη ειδική στήριξη και προσοχή. Θέλουμε να υπάρχουν λοιπόν εξειδικευμένε υπηρεσίε παροχής υποστήριξης και να μην υπάρχει δευτερογενή θυματοποίηση των θυμάτων ε, βίας βάσει του φύλου ή λόγω φύλου. Μια άλλη ιδέα για τους αστυνομικούς, τους ειδικού κτλ. Έχουμε λάβει υπόψη μας όλες τις σχετικές ε, συστάσεις και για την κατάρτιση και για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Λάβαμε πάρα πολλές προτάσεις, όλες όπως είπα τις λάβαμε υπόψη μας για να ενισχυθεί το, το δυνατόν περισσότερο αυτή η πτυχή προς όφελος των θυμάτων. Υπάρχει ένα λεπτό θέμα το οποίο αφορά τη στήριξη θυμάτων εγκληματικότητα, ιδίως ό,τι αφορά το νομικό καθεστώς, τη νομική του κατάσταση. Γνωρίζουμε ότι σε ορισμένε πολιτικές ομάδες ε, έχουν εκφραστεί ανησυχίες για τους μετανάστες που δεν έχουν δηλωθεί. Και τελικά κάποια προβλήματα που προκύπτουν με το όλο σύστημα. Εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν προσπαθούμε εδώ να αντιμετωπίσουμε την υπόθεση αυτή υποχρεώντας τα κράτη-μέλη σε ορισμένες ενέργειες ή υποχρεώνοντας να νομιμοποιήσει ε, το κάθε κράτος τους ε, αδήλωτους μετανάστες. Αλλά θέλουμε να ισχύουν τα ίδια πρότυπα με αυτά που ισχύουν και για τους δράστες, για τους θήτες. Διότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορετικοί συνδυασμοί. Δηλαδή να έχουμε ε, διδλωμένους και αδήλωτους θήτες αλλά και θύματα. Και αν τα θύματα ιδίω δεν μπορούν να αναφέρουν το περιστατικό, τότε μπορεί να μην καλύπτονται κάποια εγκλήματα, κάποιες αξιόπινες πράξεις. Άρα μπορεί να περάσουμε πλέον στο οργανωμένο έγκλημα. Ή ε, να υπάρχει έμφαση σε κάποιες συγκεκριμένες μειονότητες ή ομάδες ε, μεταναστών που θα είναι θύματα περισσότερο τέτοιων εγκληματικών πράξεων. Άλλα πράγματα τα οποία έχουμε τονίσει είναι η ανάγκη ενημέρωσης, κοινοποίηση, όταν κάποιος έχει συλληφθεί για ένα δίκημα, ανεμέρωση για το κατά πόσον έχει απελευθερωθεί ή έχει δραπετεύσει από το Σοπρανιστικό Ίδρυμα, άρνηση δικαιώματος αποκατάστασης ή αποζημίωσης. Όλα αυτά, για όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Αν το θύμα δηλαδή έχει εκφράσει επιθυμία να ενημερώνεται για αυτά, θα πρέπει αυτή η ενημέρωση να του παρέχεται. Τώρα, σε ό,τι αυτά τα το με ιδιαίτερες ειδικέ ανάγκες, Θέλουμε να υπάρχουν να είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία τα κτίρια, να υπάρχουν ειδικοί χώροι προσβάσιμοι για τέτοιου είδου θύματα, ιδίω όταν πρόκειται για περιπτώσει εκφοβισμού ή οποιασδήποτε παρενόχληση του θύματο. Τι εννοώ ακριβώ με όλα αυτά. Ε, ουσιαστικά θέλω να πω, ολοκληρώνοντα και την παρέμβασή μου, ότι Συνεργάστηκα με πολύ μεγάλη χαρά με την κυρία Χιμένεθ και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε μια πολύ καλή δέσμη συμβαστικών τροπολογιών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη σχεδόν όλες σας τις προτάσεις, οι οποίες βέβαια αυτογραμμίζονται και με τη βασική φιλοσοφία της έκθεσης. Ευχαριστώ. Thank you. Now, Senora Jiménez Ευχαριστώ, ε, κυρία Χιμένεθ Μπεσερίλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Παρμανόβα που και για μένα ήταν ιδιαίτερη χαρά να συνεργαστώ μαζί της και ελπίζω να ολοκληρώσουμε τις μας ε, με τον ίδιο τρόπο. Ε, λάβαμε, όπως υπόθηκε, περίπου 500 τροπολογίες ε, που καλύπτουν διάφορες πτυχές ε, σχετικά με τα ελάχιστα δικαιώματα. Ε, ευχαριστούμε και πραγματικά υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον από πλευρά συναδέλφων. Όπω είπε πολύ σωστά ο κ. Γκούσταυσον, πρόεδρο τη Επιτροπή Γυναικών, η πλειοψηφία των ε, τροπολογιών συμπεριλαμβάνονταν ε, στο κείμενο, απλά ενισχύουν αυτά τα οποία είχαμε γράψει. Φυσικά μας διευκόλυναν για να συντάξουμε τις συμβαστικές τροπολογίες περίπου 40 είναι αυτές, έχουν σχεδόν οριστικοποιηθεί και έλαβαν υπόψη όλα, όλες τις τροπολογίες που κατέθεσαν σχετικά με την νομική βάση, με την εφαρμογή, τους ορισμούς, τα διάφορα είδη δικαιωμάτων των θυμάτων, καθώς επίσης και την δυνατότητα των ειδικών υπηρεσιών, των εμπειρογνωμών κλπ. Ε, στόχος αυτής της εκθέσης είναι ο καθορισμός ελάχιστων κανόνων ε, σκοπός μας είναι να συντάξουμε μια οδηγία σαφή, συγκεκριμένη και κατάλληλη έτσι ώστε τα θύματα που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αισθάνονται προστατευμένα. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορούμε να πάμε πέρα από τη νομική βάση αυτής της ε, έκθεσης ή να προτείνουμε περισσότερες υποχρεώσεις για το κράτος μέλος ε, οι οποίες θα είναι δύσκολο να εφαρμοστούν στην πράξη. Στα συμβαστικέ τροπολογίε λοιπόν προθέσαμε να δημιουργήσουμε με ισορροπία ανάμεσα στις ε, ποικίλε απόψεις. Κατανοώ πω ε, η οδηγία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία πολύ σημαντική για την ε, αντιμετώπιση πολλών δικαιωμάτων και πολλών ετοιμάτων. Μιλάμε για θύματα οργανωμένου εγκλήματος, ε, βία ανάμεσα στα φύλλα, οικογενειακή βία κλπ. Θα πρέπει να επενθυμίσουμε ότι πέραν του ότι θυσιάζουμε πολλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για ελάχιστους κανόνες και εάν θελήσουμε να πάμε πολύ παραπέρα κινδυνεύουμε να μην γίνει δεκτή και έτσι να μην έχουμε ένα μέσο που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Δεν θα μιλήσω για ορισμούς, σε αυτό αναφέρθηκε η κυρία Παρμανόβα. Θα ήθελα όμως να αναφερθώ για κάποιους συνδεσμούς. Το άρθρο 1 ο στόχος ε, της, ε, για την εφαρμογή της οδηγίας και βλέπω τις ανησυχίες που εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι σχετικά με την ε, βία ε, ανάμεσα στα φύλλα. Πρόκειται για μια οδηγία η οποία εμπίπτει όμως σε ποινικέ κυρώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για μια πράξη για μια επιθετική πράξη, διότι οποιοδήποτε επιθετική πράξη που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή την έκθεση, προτιμήσαμε μια διαφορετική έκφραση, να μιλάμε για ένα ποινικό αδίκημα, που αυτό θα εγγυηθεί και την προστασία από οποιοδήποτε άλλο ε, έγκλημα που τιμωρείται ποινικά και κάναμε μια διατύπωση παρόμοια, έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα ήταν καλό, γι' αυτό και το προτείναμε. Επίσης όταν ε, τα θύματα έρχονται σε επαφή με πρώτη φορά με τις αρχές, αυτό θα πρέπει να γίνεται σε μια γλώσσα η οποία θα είναι, γίνεται κατανοητή από το θύμα. Αυτό αναφέρεται στην τροπολογία 269 και στην τροπολογία 270 πολλά θύματα βρίσκονται υπό σοκ όταν έρχονται στην επαφή αρχικά με τις αρχές σου θα πρέπει να ε, είναι απόλυτα κατανοητά τα όσα ακούνε. Εδώ αναφέρεται στην τροπολογία 135 και 136. Αναφέρεται ότι το θύμα θα πρέπει να είναι σε θέση να καταγγείλει το αδίκημα σε μια γλώσσα που κατανοεί και να έχει τις ε, ικανότητες του και, και να βρίσκεται σε, και να σε σύγχυση. Και αυτό το αναφέρουμε στην τροπολογία 280, 281, 285 και 286. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε με το Συμβούλιο είναι η σημασία να συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της οικογένειας στην οδηγία και κάτι το οποίο αντανακλάται στις τροπολογίες ε, συμπεριμένου του δικαιώματος ε, στήριξης των θυμάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 της Κομισιόν του ε, Γι' αυτό λοιπόν εγώ προτιμώ την άμεση αναφορά που γίνεται μέσω της τροπολογίας 327 ε, με ικανοποίηση δέχομαι την ε, ιδιαίτερη προσοχή που απευθύνεται στα μικρά παιδιά τα οποία είναι ε, ιδιαίτερα ευάλωτα 341 και 347 τροπολογίες πολύ Επίσης μίλησαν για την ιδέα να γίνει η ατομική αξιολόγηση κάθε θύματος. Αυτό γίνεται για να προσδιορίσουμε αν χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία το θύμα και αυτό ισχύει για όλα ε, τα θύματα, διότι κάθε θύμα είναι πρόσωπο, είναι άνθρωπος και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Κανένα θύμα δεν είναι κατώτερο από τα από τα υπόλοιπα, από όποια κοινωνική κατηγορία και αν προέρχεται. Θεωρούμε λοιπόν ότι ε, μέσα στα αδική μας θα πρέπει να συμπεριληφθούν όλα όσα αφορούν ε, εγκληματικές πράξεις, ε, λαθρεμπόριο κλπ. Συμφωνώ με την τροπολογία 448, η οποία ζητάει να υπάρχουν κάποια διαλύματα ανάμεσα στην όλη διαδικασία για τις αξιολογήσεις ε, και για να ολοκληρώσω θα θέλω να πω ότι η ατομική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τέσσερις βασικές πτυχές. Το, τα χαρακτηριστικά του θύματος, το είδος ε, του εγκλήματος, τις συνθήκες ε, του εγκλήματος και ιδιαίτερα τις επιθυμίες του θύματος. Αυτό επίσης ε, περιλαμβάνεται σε πολλές τροπολογίες. Ε, θα ήθελα επίσης να μιλήσω για την κατάρτιση των επαγγελματίων ε, τροπολογίες 199 και 200, όπως υπηρεσία, οι αστυνομίες, οι υπηρεσίες υγείας και τα δικαιώματα των, και όσων τα δικαιώματα των παιδιών. Θα πρέπει λοιπόν να θεσμοθετηθεί σε όλα τα κρατημέλη μια τέτοια κατάρτιση η οποία θα πρέπει να είναι κατάλληλη, ειδικά σε ό,τι φορά την ε, βία ε, ε, με, ανάμεσα στα φύλλα. Θα ήθελα να μάθω τι πιστεύουν οι συνάδελφοι και να μπορείτε να καταλήξουν σε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και τώρα υπό Δανική Προεδρία το Συμβούλιο έχει εκδηλώσει ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Θα θέλαμε να καταλήξουμε σύντομα το δυνατόν διότι ήδη το θέμα βρίσκεται σε καλό σημείο. Ευχαριστώ κυρία Μπεσερίλ. Θα ακούσουμε την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Αν η Κομισιόν θέλει να πει κάτι σύντομα προτού να περάσουμε στην συζήτηση. Λοιπόν, η Κομισιόν εκπροσωπείται από την κυρία Τοντίνο. Θέλετε το λέει το λόγο και Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το ε, μεγάλο ενδιαφέρον που έχει δείξει για το φάκελο αυτό. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε δει πολύ καλή έκθεση και από τις δύο εισηγήτριες, την κυρία Χιμένες και την κυρία Παρβάνοβα, καθώς και πολλές ενδιαφέρουσες τροπολογίες από άλλους ευρωβουλευτές. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για ε, στρατηγική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε εργαστεί πάνω στα θύματα εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε την απόφαση πλαίσιο από το 2001 που τώρα έχει οδηγήσει σε μια πιο ισχυρή οδηγία, πιο σαφή και με πιο σαφή περιγραφή των ε, υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των θυμάτων. Έχουμε επίσης ε, σχετική ε, ανακοίνωση του 2004. Πρόκειται λοιπόν για, την πρώτη, για το πρώτο πακέτο δικαιωμάτων των θυμάτων, το οποίο παρουσιάστηκε πέρσι και θα ακολουθηθεί και από άλλε ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος μας με την οδηγία αυτή που ήδη έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό και εφαρμόσιμο μέσο το οποίο τα κράτη-μέλη να μπορούν να το μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο ώστε να στηρίξουν τα δικαιώματα των θυμάτων ε, στις ποινικέ διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή δεν θα μιλήσουμε για τη θέση μας πάνω στις διάφορες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε όμως να επιβεβαιώσουμε ότι η προσέγγιση μας ε, πάντα ήταν οριζόντια Θεωρούσαμε ότι όλα τα θύματα θα πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία αυτή, όλες οι μορφές ε, των ε, εγκλημάτων ε, και βίαιων πράξεων, ώστε τα θύματα να έχουν το δικαίωμα να ακούγεται η φωνή τους, να προστατεύονται, να υποστηρίζονται κλπ. Ωστόσο, στην πρότασή μας αναγνωρίζουμε ότι κάποιες ομάδες θυμάτων κινδυνεύουν να υποστούν ε, περαιτέρω βλάβη κατά τη διάρκεια των ε, ποινικών διαδικασιών και γι' αυτό έχουμε συμπεριλάβει ένα κεφάλαιο για την προστασία. Όπως σας είπα δεν θα αναφερθώ στις επιμέρους τροπολογίες αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα όμως ε, να επιβεβαιώσω ότι υποστηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και το Συμβούλιο για να ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πάνω στο θέμα αυτό. Προσβλέπουμε στην ε, καλή συζήτηση πάνω στα θέματα που θύθηκαν και θα ε, υποβάλουμε συμβιβαστικές προτάσεις ώστε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο πάνω στο οποίο να μπορούν να συμφωνήσουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή. Ας ακούσουμε το Συμβούλιο, την ε, Δανέζικη Προεδρία, τον κύριο Λάρς Λίντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές και ε, τις εισηγήτριες ε, για το σημαντικό αυτό βήμα στη διαδικασία. Ε, θα έχετε ακούσει επανειλημμένα την Δανέζικη Προεδρία να λέει ότι πρόκειται για απόλυτη προτεραιότητα για την Δανέζικη Προεδρία. Είχαμε επαφές με τα κράτη-μέλη και Τολμώ να πω ότι τα δικαιώματα των θυμάτων ε, αποτελούν ε, κορυφαία προτεραιότητα, αν όχι για όλα, για, σίγουρα για πάρα πολλά από τα κράτη-μέλη. Για το λόγο αυτό η Προεδρία συμμετέχει και στη σημερινή συζήτηση. Και το γεγονός ότι φτάσατε σε αυτήν την φάση της ε, διαδικασίας μας προετοιμάζει για τους συμβιβασμούς. Καταλαβαίνουμε απόλυτα και εκτιμούμε την πολλή δουλειά που έχει γίνει για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Καταλαβαίνουμε ιδιαίτερα, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά που έχει γίνει από τις εισηγήτριες στο θέμα αυτό. Ε, φοβάμαι ότι στο εγγύς μέλλον ε, σας περιμένει ακόμα περισσότερη δουλειά. Δεν ε, ήταν μάταιη η δουλειά σας όμως. Το Συμβούλιο περιμένει να ξεκινήσει τριμερή διάλογο μαζί σας πάνω στο θέμα αυτό. Ο πρώτος τριμερής διάλογος έχει προγραμματιστεί ήδη για την επόμενη εβδομάδα. Κοιτώ τις πολύ ενδιαφέρουσες Προσλέπω στην εξέταση των τροπολογιών και τη σημερινή συζήτηση. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι υπάρχει καλή βάση για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στα θεσμικά μας όργανα με βάση κάποιες βασικές αρχές. Και ε, θα ήθελα να φέρω μερικές από αυτές. Ε, μάλιστα ε, τις ανέφεραν και οι δύο εισηγήτριες ήδη. Καταρχήν ε, το θέμα είναι ότι θέλουμε ε, οριζόντιο μέσο το οποίο να καλύπτει όλα τα θύματα εγκλημάτων συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και θα πρέπει να καλύπτουν από τα πιο ελαφρά αδικήματα μέχρι τις, ε, τα, πιο σημαντικά αδικήματα. Θέλουμε ελάχιστα επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων των θυμάτων. Εργαζόμαστε εδώ στον χώρο του ε, ποινικού δικαίου. Ε, τα θύματα λοιπόν θα πρέπει να ε, αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις ειδικέ ανάγκες τους. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε τα, οι ανάγκες ιδιαίτερα ευάλωτων ε, θυμάτων, θυμάτων με ειδικέ ανάγκες να λαμβάνονται υπόψη, αλλά το σημείο κίνησης θα πρέπει πάντα να είναι μια ατομική αξιολόγηση. Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέξουμε τις ανάγκες των θυμάτων σε διασυνοριακές περιπτώσεις ε, και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα από τα βασικά μηνύματα ε, που προέκυψε από μια πρόσφατη εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ε, υποστήριξη των θυμάτων στην Ευρώπη. Ωστόσο, δεν ε, είναι η κατάλληλη στιγμή να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Επιτρέψτε μου άλλη μία φορά να τονίσω ότι η Δανέζικη Προεδρία του Συμβουλίου δίνει μεγάλη συμφωνία στην ανοιχτή και διαφανή ε, διαδικασία διαπραγματεύσεων ε, μαζί σας και με την Επιτροπή για να πετύχουμε καλό αποτέλεσμα πάνω στο θέμα αυτό μέσα σε λογικό χρονικό διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Να ξεκινήσουμε από, τις, ε, ε, ε, από τους κοιόδους συζητητές, ο συνάδελφος ο κύριος Κροτσέτα. Να πω ότι εξετίμησα ιδιαίτερα την πρόληψη της Κομισιόν καθώς και τις εργασίες των δύο συνεισηγητριών. Ως και ο της σοσιαλδημοκρατικής ομάδας ασχολήθηκα να καταθέσω τροπολογίες ε, εκεί όπου παρατήρησα να υπάρχουν ελλείψεις ε, και όχι να προτείνω διαφορετικές θέσεις από αυτές που περιλάμβανε η έκθεση για να μην ε, δημιουργήσουμε πρόβλημα και παραφορτώσουμε μία έκθεση. Αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία θα θέλω να διευκρινίσω. Πρώτον, δεν υπάρχουν ε, αυτή την περίοδο κράτη τα οποία δεν προβλέπουν προστασία των θυμάτων εκτός αν αποκλείσουμε, αν, αν αποκλείσουμε τις ε, ολοκληρωτικές ε, χώρες όπου υπάρχουν καθεστώς χουντικό. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο έχουμε ενώπιόν μας δεν είναι τόσο το να ε, συντάξουμε μια έκθεση η οποία ε, ήδη καλύπτεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή από την ε, διεθνή νομοθεσία. Αλλά να συμπεριλάβουμε κάποια καινοτόμα στοιχεία μπορούν να προστατεύσουν τα θύματα που αυτή τη στιγμή σε κάποια κράτη δεν προστατεύονται ή και να καταλήξουμε στον ορισμό του όρου θύματος. Εάν ένας ε, έμπορος ναρκωτικών ε, χάσει τη ζωή του καρδιάρκεια μιας ανταλλαγής ε, ε, πυροβολισμών με έναν συνάδελφό του μαφιόζο, τότε θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση. Αν ένας μαφιόζος χάσει τη ζωή του τη στιγμή που μάχεται για την ε, απόκτηση ενός, ε, μιας περιοχής, ε, για τον έλεγχο μιας περιοχής, τότε αυτό δεν μας αφορά. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τα αθώα θύματα, διότι εκεί είναι που το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει την προστασία του πολίτη, του αθώου. είναι νοικοκυρά λοιπόν ή τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο στην Τουλούζη και δολοφονούνται είναι αθώα θύματα. Ο τρομοκράτης όμως ε, που προσπαθεί να σκοτώσει και χάνει τη ζωή του δεν είναι αυτό θύμα, δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη προστασία. Έχει την προστασία ή ουδήποτε ανθρώπου κατά την διάρκεια μιας δίκης εάν και εφόσον εμπλακεί σε μια τέτοια περιπέτεια αλλά και τίποτα παραπάνω. Η τροπολογία μου λοιπόν αυτό ήθελε να διευκρινίσει. Δύο άλλα ζητήματα και ολοκληρώνω. Ε, στην ποινική δικονομία για να θεωρηθεί ένας άνθρωπος θύμα θα πρέπει να πέσει θύμα ενός αδικήματος. Αλλά αν για λόγους ε, φιλετικούς ε, ηθαγένειας ε, ζει σε μια κατάσταση μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πρόσωπο ως θύμα πέραν πέραν της καταστάσεως ε, της εξευθελιστικής στην οποία ζούσε και συνεχίζει να ζει. Λοιπόν, να λάβουμε υπόψη του ε, άστεγους οι οποίοι μπορούν να ε, φυλακιστούν επειδή δεν έχουν κάποιο, κάποια στέγη πάνω το κεφάλι τους και ζουν στο δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να προσδιορίσουμε και το καθεστώς του θύματος που δεν ε, σχετίζεται πάντα με την διάπραξη ενός αδικήματος. Μερικές φορές υπάρχουν, όπως παραδείγματος χάρη στις χώρες που ε, δεν, ε, μάλλον που τιμωρούν τους ομοφιλόφιλους ε, ή δεν τους παρέχουν τα δικαιώματά τους και κάτι ακόμα. Ο Σάλμα Ανδράσουντι που ζει στην, <clears throat> στον Βασίλειο εδώ και 20 χρόνια διότι έχει πέσει θύμα μιας φάτβα που από πλευράς ε, των ε, Ισλαμιστών των φαρατικών είναι θύμα ή δεν είναι θύμα. Σύμφωνα με την νομοθεσία δεν είναι θύμα διότι δεν έχει διαπραχθεί κανένα έγκλημα. Αλλά αυτός ο κύριος μένει σε ένα μπούνκερ εδώ και 20 χρόνια και δεν έχει το δικαίωμα ακόμα και αν υπάρχει μία διαδικασία ενώπιον ε, δικαστηρίου για ενάντια των ε, ατόμων που έχουν εκδώσει αυτή τη βάτβα. Θα σας αναφέρω και τον ε, Σαβιάνο, ο Ρομπέρτο Σαβιάνο λοιπόν, που έχει καταδικαστεί σε θάνατο από την Ναπολιτανική Καμόρα, δεν είναι θύμα και δεν μπορεί να συμμετέχει στην Ιταλία σε καμία δίκη, ακόμα και αν γνωρίζουμε αυτούς που επιθυμούν να, τον δολοφονήσουν, διότι δεν έχει πέσει θύμα. Το λέω αυτό στις ηγήτριες. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει ιδιαιτερότητα να είναι κάποιος να απειλείται μάλλον κάποιος από τρομοκράτες ή από τη μαφία από... είναι διαφορετικό από το να απειλείται από τον γείτονά του, διότι η αστυνομία μπορεί να τον ελέγχει αυτόν. Αλλά αν το, όταν το ενδυνάμει θύμα έχει καταδικαστεί από τρομοκρατικές ε, οργανώσεις ή από άλλες εγκληματικές διεθνείς οργανώσεις, ποιος μπορεί να υπερασπιστεί αυτά τα άτομα. Θεωρώ λοιπόν ότι λίγο περισσότερο κουράγιο Δηλαδή να πάμε πέραν της ισχύψας τάξης και να ε, προτείνουμε ένα νέο σχέδιο διότι η Ευρώπη δεν ε, πρέπει να κάνει τον ε, ταμεία των νομοθεσιών και να καταλήγει μετά σε συμβασμούς. Η Ευρώπη έχει νόημα εάν προωθήσει μια μεγάλη δημοκρατική και φιλελεύθερη επανάσταση και να οδηγήσει τα κράτη τα οποία ε, έχουν επιφυλάξει να προχωρήσουν. Αν κατορθώσουμε λοιπόν σε αυτό το έργο μας ε, θα είμαστε χρήσιμοι. Διαφορετικά δεν κάνουμε τίποτα άλλο που να επαναλαμβάνουμε τις εργασίες των Εθνικών Κοινοβουλίων. το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τρία θέλω πράγματα να πω. Πρώτα απ' όλα να επιστρέψω την προσοχή σας σε μία ενημέρωση από το Library για θύματα περιβαλλοντικών εγκλημάτων. Το να είναι κάποιο θύμα περιβαλλοντικού εγκλήματο, ή μελλοντικέ γενιέ να είναι θύμα περιβαλλοντικού εγκλήματο, πιστεύουμε ότι είναι κάτι που πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτήν την οδηγία. Έχουμε καταθέσει δε δύο τροπολογίε, 207 και 227 συγκεκριμένα. Σε αυτές λέμε ότι το περιβαλλοντικό έγκλημα δεν είναι λιγότερο έγκλημα από άλλα. Μπορεί να μην έχουμε ένα θύμα ε, που μπορεί κανείς να το δει εύκολα, αλλά μπορεί να πρόκειται για έγκλημα προς ε, τη σε βάρο της επόμενη γενιάς. Το περιβάλλον δηλαδή ουσιαστικά είναι το θύμα σε αυτή την περίπτωση. Και θα πρέπει να το δούμε αυτό. Άκουσα τι λέει και ο κύριος Κροτσέτα άνοιξε τη συζήτηση ποιος είναι θύμα ποιου πράγματος. Εγώ παραμένω εντός της οδηγίας. Θύματα εγκλημάτων. Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα είναι και αυτά εγκλήματα. Ποιο είναι θύμα ενό περιβαλλοντικού εγκλήματο, λοιπόν, ιδού η απορία. Πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο. Το θύμα, το αντιμετωπίσμα ω θύμα ενό συγκεκριμένου εγκλήματο. που οδηγεί σε ανάγκη προστασίας. Ένα θύμα είναι πιο ευάλωτο λόγω του εγκλήματος το οποίο έχει διαπραχθεί ή λόγω των προσωπικών του χαρακτηριστικών. Και το προσωπικό χαρακτηριστικό τελικά είναι κάτι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη ως κάτι που κάνει έναν άνθρωπο πιο ευάλωτο Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει πράγματι η ατομική αξιολόγηση. Συμφωνούμε απόλυτα. Το λένε και δύο εισηγήτριε και αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο τη όλη οδηγία. Αν λοιπόν έχουμε μια καλή ατομική αξιολόγηση, πολλά άλλα πράγματα, πολλοί ορισμοί για το τι καθιστά κάποιον πιο ευάλωτο, αν αυτό είναι το έγκλημα ή αν είναι κάποιο προσωπικό χαρακτηριστικό, δεν θα είναι πλέον και τόσο σκόπιμα. Έχουμε και την τροπολογία 162 όμως, όπου εκεί τι λέμε, Μιλάμε για άτομα χωρίς ε, νόμιμα χαρτιά, αδήλωτους, ε, μετανάστες, που μπορεί να είναι θύματα και δεν έχουν χαρτιά. Αυτό αλλάζει κάτι, δεν είναι θύματα. Και στο πλαίσιο της δικαστικής εξέτασης περίπτωσής τους και πιο πέρα, πρέπει και αυτό να λαμβάνεται υπόψη. τα δικαιώματα των αδήλωτων ε, μεταναστών, ίσως να είναι κάτι που δεν θέλει κανείς να το θίξει εύκολα. Αλλά γιατί να μην αρχίσουμε με τον ορισμό του εγκλήματος και όχι με τον ορισμό των προσωπικών χαρακτηριστικών. Κανένα θύμα δεν είναι λιγότερο θύμα από κάποιο άλλο. Αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη θέση των προσφύγων και μεταναστών. και να καταλήξουμε σε πολλούς αφισορισμούς για να αποφύγουμε την περαιτέρω θυματοποίηση. Δηλαδή να ξαναγίνει θύμα το θύμα. Θύμα του ίδιου εγκλήματος για δεύτερη φορά. Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε να παθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ε, υπάρξει θύματα τρομοκρατικής ενέργειας ή οργανωμένου εγκλήματος. Βέβαια, μπορούμε να είμαστε τόσο αυστηροί σε αυτή τη διατύπωση. αθώα θύματα ή θύματα εν γέννη. Πάντω το κύριο Κροτσέτα εδώ πέρα. Μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να ορίσουμε τι είναι αθώο και τι δεν είναι αθώο θύμα. Μία γυναίκα θύμα σωματεμπορίας, διακίνησης, που μπορεί και να το ξέρε κιόλα. Για να εκπορνευθεί, την ε, ε, χρησιμοποίησαν, τη διακίνησαν. Είναι αθώα ή δεν είναι αθώα τελικά δεν αξίζει προστασία επειδή μπορεί να γνώριζε, δεν είναι αθώα. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοια διάκριση. Εντάξει, έχετε κάποια πιο συγκεκριμένα παραδείγματα για την τρομοκρατία και για τα οργανωμένα εγκλήματα. Α, εδώ μιλάμε για πράγματα που οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι και τόσο σαφείς. Τρίτον και τελευταίον, βιαζόμαστε τόσο πολύ και έρχομαι στο Συμβούλιο. Την επόμενη εβδομάδα Έχουμε ψηφοφορία. Έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό νομοθέτημα στα χέρια μας. Δεν νομίζω ότι βιαζόμαστε. Από τη στιγμή που εξακολουθούμε να συζητάμε τι θα πει θύμα, τι δικαιώματα θα πρέπει να έχει, ποιος είναι θύμα, ποιος δεν είναι κτλ. Είπα και αυτό για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα. Να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Νομίζω ότι παραβιαζόμαστε. Θέλουμε να πετύχουμε συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Μα δεν θα έχουμε δώσει μια καλή εντολή στους διαπραγματευτές μας, δεν θα δίνει ξεκάθαρη εντολή. Και αν οι διαπραγματευτές μας δεν έχουν ξεκάθαρη εντολή, δεν θα είναι και καλό το αποτέλεσμα. Ή δεν θα είναι σαφές τέλο πάντων. Συμφωνώ ότι ναι πράγματι, εδώ και κάποιο χρόνο είναι έτοιμο το Συμβούλιο, λένε και οι συγγύτρε, ωραία να βιαστούμε κι εμείς. Όχι, δεν συμφωνώ. Για άλλα θέματα, για τους πρόσφυγες, να αναφέρω το Δουβλίνο. Δεν βιάζεται το Συμβούλιο εκεί πέρα και το περιμένουμε. Γιατί να μας περιμένει και αυτό τώρα. Η εντολή καταρτίστηκε επί Πολωνικής Προεδρία. Τώρα είμαστε στη Δανική Προεδρία. Αλλάζει άποψη. Και αν ναι, δεν πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μάκιντάιρ, έχετε σειρά εσείς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που ο Τίμωθη Κέρκοπο και ο εισηγητή δεν είναι εδώ. Θα έπρεπε αυτό κανονικά να μιλά στη θέση μου, αλλά έχω την ε, δήλωσή του μπροστά μου. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τι δύο για το έργο του. Και να πω ότι η ομάδα μου στηρίζει απόλυτα τους στόχους της έκθεσης αυτής. Έχω δύο-τρία σχόλια. Προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο και είμαι ιδιαίτερο υπερήφανη για το ότι η Επίτροπο Ρέντινγκ μίλησε για τι βέλτιστε πρακτικέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Για μια φορά τουλάχιστον ε, κάποιος μας αναφέρει ω του καλούς τη υπόθεση. Όμως έχω μια ανησυχία. Καταρχά γιατί επεκτείνουμε τόσο πολύ την έκθεση, ώστε τελικά να κολλήσει στο Συμβούλιο και να μην ε, ευημερήσει τελικά ενδεχομένω, να μην ευοδοθεί αυτή η έκθεση. Ας μείνουμε λοιπόν στου τομείς που καλύπτει η έκθεση και ας μην περάσουμε σε τομείς όπως είναι το περιβαλλοντικό έγκλημα, όπου εκεί όλοι είναι θύμα τελικά. Ένα άλλο πρόβλημα που έχω είναι η διάκριση μεταξύ αθώων και μη αθώων θυμάτων. Πριν δικαστεί κάποιο στο δικαστήριο και καταδικαστεί, είναι αθώος. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Ακόμη και αν μπορεί να πιστεύουμε ότι είναι τρομοκράτης ή οτιδήποτε άλλο. Η αθότητα δεν είναι η γνώμη κάποιου. Είναι θέμα που αποφασίζει ένα δικαστήριο. Άρα είναι επικίνδυνο να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Κάτι άλλο που με ανησυχεί είναι ότι δημιουργούμε πάρα πολλά ειδικά θύματα Και για να είμαι ειλικρινής, οποιοδήποτε ήταν θύμα τρομοκρατικής ενέργειας, κάποιου εγκλήματος τύπου μαφίας, βιασμού, σεξουαλικής κακοποίησης κτλ. Έχουν περάσει φρικτές στιγμές. Και όλοι αξίζουν την κατηγορία θύμα να ενταχθούν σε αυτήν την κατηγορία. Είναι ανησυχητικό το ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιεράρχηση θυμάτων, όπου άλλα θύματα είναι πιο σημαντικά από κάποια άλλα. Με ανησυχία αυτό λοιπόν. Αμφισβητούμε και κάτι ακόμη. Μπορεί και να είμαστε σε μια... Ε, μπορεί να κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε δικαιώματα. Αλλά στερούμε τα θύματα του δικαιώματος που έχουν ουσιαστικά. Δηλαδή την καταδίκη του εγκληματία. Να δουν να καταδικάζεται ο δράστης. Αυτό είναι το βασικό δικαίωμα. Ναι, φυσικά και το θύμα πρέπει να έχει ευελιξία για τι συνεντέξει, για τι ακροάσει, για την παρουσία του στο δικαστήριο. Ε, μπορεί να θεωρούν τα θύματα ότι αυτό είναι προ όφελό του, αλλά μπορεί τελικά να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η δίκη ή να τη γλιτώσει ο δράστη. Μήπως ε, τελικά συγχαίρουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δικαίωμα και αυτό που θέλουν ουσιαστικά τα θύματα, δηλαδή να καταδικαστεί ο δράστης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν ρεαλιστέ. Αυτό έχει αναφέρει και η Δανική Προεδρία. Αν λοιπόν υπερβούμε το πεδίο εφαρμογή οδηγία αυτής, νομίζω ότι θα πάμε πουθενά. Θα καταλήξει στο κενό Έχω λοιπόν αυτές, αυτούς τους περιορισμούς και αυτές τις επιφυλάξεις. Κατά τα άλλα εγκρίνω την έκθεση. Πρόεδρος, δεν βλέπω να σηκώνει κάποιος άλλος να άλλο στο χέρι. Οπότε μπορούμε να επανέλθουμε στις, ε, ε, στον συμπρόεδρο καταρχάς, τον κύριο Γκούσταυσον και μετά στις δύο εισηγήτρες. Ναι, θα Ήθελα να πάρω το λόγο περισσότερο ως όδης συγητής ε, παρά ως ε, συμπρόεδρος. Θα είμαι σύντομος. Όπως είπα νωρίτερα, οι, ε, οι συγγήτριες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και έχουν συμπεριλάβει πολλά καλά θέματα και στηρίζω απόλυτα τις 40 συμβιβαστικές τροπολογίες, εκτός από δύο. Ήθελα να να τονίσω ένα σημαντικό θέμα, τον ορισμό ε, της ε, βίας του φύλου. Μιλάμε για ε, βία ανδρών κατά των γυναικών. Μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι σημασιολογικό το θέμα, ότι δεν έχει πολύ σημασία. Όταν όμως ε, μιλάμε για βία ε, σε στενές σχέσεις, ναι, υπάρχει βία γυναικών κατά των ανδρών, υπάρχει και βία σε ομόφιλες σχέσεις, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό, το 90% ε, της βίας, είναι βία ε, ανδρών κατά των γυναικών και αυτό θα πρέπει να τονίσουμε. Αλλιώς προσπαθούμε να κρύψουμε τον, ε, την πατριαρχική δομή στην κοινωνία μας. Υπάρχει μια έννοια που χρησιμοποιείται και σε διεθνές επίπεδο και σε διάφορα πλαίσια έχει υιοθετηθεί από ε, όλα τα κράτη-μέλη και συμπεριλαμβάνεται και στο, στην πλατφόρμα του, του Πεκίνου ε, χρησιμοποιείται η βία ανδρών εις βάρος των γυναικών. Ε, αλλά είναι σημαντικό να αποφύγουμε ε, αυτή την έκφραση διότι οποια, οποιαδήποτε άλλη βία η πράξη ε, είναι εξίσου σημαντική στις στενές σχέσεις μεταξύ ανθρώπων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να βρούμε άλλη διατύπωση. Αλλά όπως είπα είναι εξαιρετική δουλειά και στηρίζω τη ε, δουλειά των δύο εισηγητριών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκούσταυσον. Αν ε, δεν ε, υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, να απευθυνθούμε και πάλι στις εισηγήτριες για να κλείσουμε τη συζήτηση. Να ακολουθήσουμε την ίδια σειρά με την αρχή. Να δώσουμε πρώτο το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις ε, παρατηρήσεις ε, του κυρίου Κροτσέτε, ε, Κροτσέτα, είναι ακριβώς αυτή η προσέγγιση μας. Προσπαθούμε να βρούμε νέους τρόπους να αντιμετωπίσουμε τα θύματα και να κάνουμε την πορεία μέσα από το σύστημα πιο εύκολη για, αυτό, για αυτούς. Έχουμε καταβάλει πολλές προσπάθειες για να τους ε, καλύπτουμε όχι μόνο, ε, ε, να στηρίζουμε όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά να έχουν τις σωστές πληροφορίες, να ξέρουν πού πρέπει να πάνε και να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει μαζί τους και όχι να εξισώνονται με τον με τον δράστη στο τέλος της διαδικασίας, κάτι που συχνά συμβαίνει. Έχουμε την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που λέει ότι διάφορες ομάδες ε, θυμάτων αποτελούν ε, αντικείμενο στιγματισμού από το σύστημα και γι' αυτό προσπαθούμε να τους δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Όσον αφορά την έννοια του θύματος, νομίζω ότι αυτή προέρχεται από το πρωτογενές δίκαιο. Ε, και από τη βασική αρχή ότι ο καθένας είναι αθώος ε, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες όμως, ε, διότι είναι μάλλον ηθικό και όχι τόσο νομοθετικό το θέμα. Όσον αφορά αυτά που είπε η κυρία Σαρτζεντίνη και τις προτάσεις της, τα θύματα περιβαλλοντικού εγκλήματος, έχουμε συζητήσει το θέμα, διότι μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο συνολικός πληθυσμός ενός χωριού, για παράδειγμα, μπορεί να αποτελεί θύμα ε, περιβαλλοντικού εγκλήματος ή κάποιου ατυχήματος. Ε, όσον αφορά όμως σε την νομοθεσία που καλύπτει τα περιβαλλοντικά ατυχήματα και άλλα ε, θέματα που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στον πληθυσμό, δεν νομίζω ότι είναι εδώ το κατάλληλο σημείο να αναπτύξουμε την ιδέα των θυμάτων του περιβαλλοντικού εγκλήματος. Όσον αφορά τα θύματα με συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κατηγορίες, προσπαθούμε να ε, εισάγουμε την έννοια της ατομικής αξιολόγησης, απαντώ και στην κυρία Μάκιντάιρ. Και γι' αυτό καταβάλαμε κάθε προσπάθεια να έχουμε τέσσερα σαφή κριτήρια ε, προσωπικά χαρακτηριστικά, τύπο του εγκλήματος ε, και την θέση του θύματος και έχουμε ε, δώσει το μέσο αυτό στα κράτη-μέλη για να κάνουν την ατομική αξιολόγηση αντί να χωρίζουμε τον κόσμο σε διάφορες κατηγορίες στην οδηγία αυτή. Συμφωνώ επίσης απόλυτα ότι οι μετανάστες, ε, ε, οι μετανάστες χωρίς επίσημα έγγραφα και οι πρόσφυγες άσχετα από το νομικό τους καθεστώς είναι άνθρωποι στους οποίους ε, θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των θυμάτων. Ιδιαίτερα αν είναι δράστες είναι σημαντικό να έχουν πλήρη κάλυψη όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, παραβατών. Δεν καταλαβαίνω γιατί λοιπόν να ισχύει κάτι διαφορετικό ε, για τα θύματα. Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, όταν ξεκινήσαμε τις εργασίες πάνω στην πρόταση αυτή, αρχικά, κατά την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, ανακοινώσαμε το χρονοδιάγραμμα, καθώς και κατά την παρουσίαση του Σχεδίο έκθεσης και κατά την ανταλλαγή απόψεων με τους κοιόδης εισηγητές ε, κατά την τελευταία σύνοδο του Στρασβούργου. Ε, το χρονοδιάγραμμα το προτείναμε λοιπόν ήδη από την αρχή και διαμορφώθηκε έτσι όχι επειδή είναι έτοιμο το Συμβούλιο αλλά επειδή υπάρχει ισχυρή πίεση από κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις οι οποίες ασχολούνται με το θέμα της ε, βίας ε, εξαιτίας του φύλου. Υποσχεθήκαμε λοιπόν ότι ε, χωρίς καθυστέρηση θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οδηγία που να καλύπτει τα δικαιώματα των θυμάτων. Επίσης όσον αφορά τα ε, θέματα που ανέφερε ο κύριος Γκούσταυσον. Ε, καθ' όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων προσπαθήσαμε να βρούμε μια, έναν καλό συμβασμό όσον αφορά ε, το, την ε, βία εξαιτία ε, του φίλου Ε, και συνήθως οι γυναίκες ε, είναι θύματα τέτοιων εγκλημάτων και ο ορισμός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι κάπως περιορισμένος, διότι καλύπτει ε, μόνο ε, την βία εξαιτία φύλου εις βάρος γυναικών και δεν καλύπτει όλες τις άλλες πτυχές, ε, δεν καλύπτει για παράδειγμα... άτομα που ανήκουν στην κατηγορία ΛΟΑΔ, ε, λεσβείες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι και διεμφυλικοί. Το θέμα λοιπόν ε, είναι να μην καλύψουμε μόνο το, τη βία εις βάρος των γυναικών, αλλά όλα τα θύματα. Γι' αυτό η βασική μας προσέγγιση θα πρέπει να είναι να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλα τα θύματα, να είμαστε ουδέτεροι ως προς το φύλλο και κατόπιν να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα των γυναικών. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τους δύο αυτούς ορισμούς, ε, την βία εξαιτίας ε, φύλου και την βία σε στενές σχέσεις. Ε, και κατόπιν ε, με τα εκτιμώντας προσπαθούμε στο βαθμό που είναι δυνατόν να καλύψουμε το θέμα αυτό. Ε, πάντως ε, μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας κατά τη διάρκεια των συμβαστικών προτάσεων, τροπολογιών. Και καταλαβαίνω ότι ω πρόεδρο τη Επιτροπή Γυναικών ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό, πάντω θα το συζητήσουμε. Κυρία να πω στον κύριο Κροτσέτα πως ε, συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενά του και πως ήθηκα, ήθηκα το τονίζω, ένας τρομοκράτης ο οποίος ε, κουβαλάει μία βόμβα για να φωνεύσει και κρύγνεται στα χέρια του δεν ε, είναι το ίδιο πράγμα με ένα παιδί το οποίο θα σκοτωνόταν εάν έσκαγε η βόμβα. Χαίρομαι που το λέτε και εγώ το επιβεβαιώνω. Ο Σάλμα Ράσοντε είναι θύμα, είναι θύμα της τρομοκρατίας. Δεν ξορίζουμε ε, πώς ε, θα προστατευτεί διότι η απειλή έρχεται, μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι μια οδηγία που δεν πάει πολύ μακριά, αλλά μπορώ να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε προκειμένου να υπάρξει και μια άλλη οδηγία, ένα άλλο είδου οδηγία που πράγματι θα λαμβάνει υπόψη και θα προστατεύει αυτό τα δικαιώματα που εσεί εσείς αναφέρατε. Τούτου λεχθέντος εσείς ε, λέτε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν μια πολύ αποτελεσματική νομοθεσία από τι άλλες. Να σας πω ότι όλες οι οργανώσεις ε, θυμάτων, στήριξη των θυμάτων και τα θύματα που ήρθαν ε, από την ε, Σκοτία, Ελλάδα κλπ. Λένε ότι μια γυναίκα που βιάστηκε σε μια ξένη χώρα για το παιδί της το οποίο α, Πιστεύω λοιπόν πως ε, αυτή η οδηγία θέλει να προσφέρει προστασία και υποστήριξη στα άτομα τόσο επίπεδο μετάφρασης, διερμηνίας, ε, προστασίας, ε, μάλλον ε, στήριξης ε, των οικείων σε περίπτωση θανάτου. Η αστυνομία αναγνωρίζει τι πρέπει να κάνει, οι δικαστές επίσης, σε όλα αυτά όμως απάντη, απαντήσαμε προηγούμενα. Πιστεύω λοιπόν ότι κάναμε καλή δουλειά, αδιάκοπα δουλέψαμε, το λέω για τη Γραμματεία, για την Κομισιόν, για το Συμβούλιο, για όλους μας εδώ στο Κοινοβούλιο το γνωρίζαμε από τον Ιανουάριο το χρονοδιάγραμμα και οι σκιώδεις εισηγητές συνεδριάσαμε επανειλημμένα. Εγώ λοιπόν ε, επιθυμώ να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα, να περάσουμε στον τριμερή διάλογο που δεν θα είναι κάτι το εύκολο και το απλό. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε των επιθυμιών μας και από τον κύριο Κροτσέτα και σε όλους όσοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου είμαι πρόθυμη προκειμένου να βελτιώσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μήνυμα ελήφθη. Ε, ακούσαμε την άποψη που εξέφρασαν και οι δύο συγγήτριες αυτό τον τόσο ευαίσθητο ζήτημα και η ψηφοφορία θα πρέπει να ε, λάβει χώρα όσο νούπο, Μάρτιο 27 συγκεκριμένα. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. 27 θα ψηφίσουμε λοιπόν. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών που ήρθαν σήμερα ανάμεσά μας. Τώρα Συνεχίζουμε ακάθεκτη στο επόμενο σημείο της Μεσσίας Διατάξεως. Άκουσα στις 28, μάλλον δεν άκουσα καλά πρόεδρε, ναι, 27, 27. Ευχαριστώ. 27 Μαρτίου. I see, I see. I have been reported that although, although the rapporteur... Μολονότι ότι η κυρία Βέμπερ είναι παρούσα ήδη και επειδή η Κομισιόν θα πρέπει να λάβει μέρος στην συζήτηση, δεν έχει φτάσει ακόμα, έχει καθυστερήσει. Μια πολύ σύντομη διακοπή 20 λεπτών 16 και, 16 και 40, 16 και 44 και 40 λοιπόν θα ξεκινήσουμε το επόμενο σημείο. Thank you for your attention. Thank you for your attention. That's good. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να συνεχίσουμε με το σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης. Το σημείο αυτό αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 562 με σκοπό τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά με την προσωρινή επαναφορά του ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικέ περιστάσει. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Ρενάτε Βέμπερ. Έχουμε λοιπόν εδώ την εξέταση των τροπολογιών. 80 τον αριθμό. Ναι. Ούτε λιγότερε ούτε περισσότερες. Η εισηγήτρια σήμερα θα μας παρουσιάσει τα κύρια στοιχεία των τροπολογιών για να δούμε πώς μπορεί να ρυθμιστεί η ενδεχόμενη επαναφορά ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα λεπτό πολιτικό ζήτημα. Θα ακούσουμε πρώτα την εισηγήτριά μα και μετά θα ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπο ή εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Μόνικα Μό μοσχαμερ δεν έχει έρθει ακόμη. Αλλά α δώσω το λόγο στην συνάδελφό μα Ρενάτε Βέμπερ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου που κατέθεσαν τροπολογίες για την έκθεση αυτή. να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους συναδέλφους που μου έγραψαν μηνύματα για να μου εξηγήσουν ε, τις απόψεις τους. Το εκτίμησα ιδιαίτερα. Επίσης εκτιμώ το γεγονός και κατανοώ ότι για διάφορους λόγους κάποιοι συνάδελφοι έχουν διαφορετικές απόψεις για κάποιες από τις δικές μου προσεγγίσεις στην έκθεση αυτή. Σε αυτό το στάδιο θα προτιμούσα να σας παρουσιάσω τις δικές μου τροπολογίες στην έκθεση. Είχα πολύ καλή συνεργασία με τον συνάδελφο Έντζο από την ομάδα των Σοσιαλιστών για την σύνταξη και κατάθεση των τροπολογιών. Θα σας εξηγήσω γιατί θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να καταθέσουμε αυτές τις τροπολογίες και πρώτα απ' όλα θέλω να τονίσω ότι ήθελα να εξασφαλιστεί ότι υπό καμία συνθήκη σε όλο το κείμενο ε, ήθελα να πω ότι οι μεταναστευτικές ροές, η διέλευση των συνόρων από μεγάλο ρυθμό ανθρώπων σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί να χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο για την επανεισαγωγή δηλαδή ελέγχων στα σύνορα. Έχω καταθέσει και σειρά τροπολογιών για το θέμα αυτό. Διαδικασία επιστροφής. Είναι ένα άλλο θέμα το οποίο αναφέρεται σε κάποια άρθρα. Γιατί αυτές οι διαδικασίες ουσιαστικά δεν είναι στα χέρια των κρατών μελών. 100%. Εξαρτώνται και από τη θέση της τρίτης χώρας. Μια άλλη θέση μετροπολογιών αναφέρεται στην ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας της όλης διαδικασίας που προτείνουν. Στο άρθρο 24, παράγραφος 3 και παράγραφος 4 γίνεται λόγος για την ε, δημοσίευση γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μετά μιλάμε για τη διεξαγωγή κοινών συναντήσεων. Να μην είναι αυτά υποχρεωτικά ε, βήματα στο πλαίσιο της διαδικασίας, αλλά εάν χρειαστεί, if necessary, να προσθεθεί αυτή η φράση. Δηλαδή, αν τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται να δημοσιεύσει κάποια έκθεση κομισιών. Το ίδιο ισχύει για τις κοινέ αυτές συναντήσεις των κρατών μελών που έχουν υπανεισαγά για τους ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Να έχουν δηλαδή συναντήσεις με τα αλλα κρατημέλη και με την Κομισιόν. Και αυτό να είναι το δηλαδή αν χρειάζεται να γίνεται. Σε ό,τι αφορά την έκδοση κατευθυντηρίων γραμμών από την Κομισιόν, μιλάω πάντα στο πληθυντικό γιατί όπως προείπα, είναι τροπολογίες κοινέ που κατέθεσε ο κύριος ε, Έντσου και εγώ. Λοιπόν, σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά στην προηγούμενη εμπειρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την επανεισαγωγή ελέγχων στα σύνορα. Ο εκπρόσωπος ή η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε είχε αναφέρει ότι είναι δύσκολο για την Κομισιόν να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές ή να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές. Αλλά θεωρήσαμε ότι μπορεί κάτι να γίνει από την Κομισιόν, γιατί τελικά η Κομισιόν στη δική της πρόταση ζητούσε να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τα θέματα της επαναφοράς έλεγχο στα σύνορα. Αν είναι έτσι λοιπόν τα πράγματα, που μάλλον είναι, τότε η Κομισιόν κάτι μπορεί να κάνει. Άρθρο 26. Να αποφασίζει δηλαδή η Κομισιόν για την επαναφορά των ελέγχων αφού μελετήσει αντελεχώς την κατάσταση αν θυμάμαι καλά και αν θυμούνται και οι συνάδελφοι καλά, είχε γίνει μια συζήτηση και είχαμε πει ότι πρέπει να αναφέρεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Ε, άρα πήραμε ως απόφαση να αναφέρουμε την ε, επιτροπολογία, αλλά να ζητήσουμε να είναι πιο διαφανή σε όλη η διαδικασία. Έτσι, θα υπάρχει ταυτόχρονα δυνατότητα και να γίνει συζήτηση και μετά να μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει τις αποφάσεις. I considered that no extra conditions Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμπεριφθούν προϋποθέσεις, αφού γίνει δηλαδή αξιολόγηση της κατάστασης ένα κράτος μέλος. Και αν θέλουμε παραπάνω πράγματα, δηλαδή να εντοπιστούν ενδεχόμενες απειλές προς τη δημόσια ασφάλεια στην εσωτερική πολιτική. Αυτό θα καταστήσει μια αποτελεσματική τη διαδικασία. Και μπορεί κανείς να διορθωθεί πότε τελικά θα είναι η Κομισιόν σε θέση να λάβει μια απόφαση. Άρα δεν θέλουμε να μπουν αυτοί επιπλέον. Αυτές οι επιπλέον παράμετροι. Τώρα τέλο ό,τι αφορά το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει μια τροπολογία η οποία ζητά από την Κομισιόν να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τουλάχιστον σε αιτήσια βάση μία έκθεση. Φυσικά, μακάρι, αν χρειάζεται, η Κομισιόν να υποβάλει περισσότερες της μιας εκθέσεις αν έχει υπάρξει πάνω φορά ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε περισσότερες της μιας περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τι άλλες τροπολογίες, τροπολογίες που κατέθεσαν οι συνάδελφοί μου, νομίζω ότι μπορούμε να τι ομοδοποιήσουμε σε αρκετές κατηγορίες. Μια δέσμη τροπολογιών είναι από συναδέλφου που δεν επιθυμούν καμία αλλαγή στην ε, ισχύουσα κατάσταση. που δεν τους αρέσει και τόσο ο χώρος του Σέγγεν. Υπάρχουν άλλες τροπολογίες που δίνουν έμφαση στο ρόλο του κράτους μέλους, σε αντιδιαστολή με το ρόλο της Κομισιόν. Υπάρχουν επίσης τροπολογίες που σε κάποιο βαθμό ευθυγραμμίζονται με την έκθεση που έχω καταρτήσει αλλά φυσικά θα ακούσω με τα χαρά και τα επιχείρηματα των συναδέλφων. Εγώ έχω καταλήξει σε αρκετές συμβαστικές τροπολογίες που πιστεύω ότι μπορούμε να συντάξουμε. Αφού βέβαια συνεργαστούμε, αφού έχουμε κάποιες ακόμη συναντήσεις μεταξύ μας και συζητήσουμε όλες αυτές τις τροπολογίες, αλλά φυσικά και το πρωτότυπο, το αρχικό κείμενο. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ για τώρα. Να ακούσω τι θέλει να μας πει το Συμβούλιο ενδεχομένω η Κομισιόν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Okay, how about the commission or the... Ωραία. Θέλει να παρέμβει η Κομισιόν ή ε, το Συμβούλιο. Παρακαλώ, η κυρία Μοσχάμερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, σας ευχαριστήσω για όλες τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν και να κάνω μία γενική παρατήρηση. Υπάρχουν αρκετές τροπολογίες που τονίζουν την σημασία της ε, επανεισαγωγής ως έσχατη λύση. Ε, μερικές τροπολογίες είναι ίσως ε, κάπως υπερβολικές. Θα ήθελα να επανέλθω και στην τροπολογία για τις κατευθυντήριες ε, γραμμές όσον αφορά τις ε, απειλές, ε, εθνικής πολιτικής, τις απειλές προς την εθνική πολιτική ή για λόγους ασφαλείας. Έχουμε κάποιες ανησυχίες για το θέμα αυτό, διότι πρέπει να κοιτάξουμε τα θέματα αυτά κατά περίπτωση. Είναι αλήθεια ότι η Επιτροπή στο τέλος ε, λαμβάνει την απόφαση. Παρ' όλα αυτά η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη μέσω της ε, λεγόμενης διαδικασίας της επιτροπολογίας. Ε, συμμετέχουν λοιπόν απόλυτα τα κράτη-μέλη και μας ενδιαφέρει πολύ η θέση των κρατών μελών. Όσον αφορά το άρθρο 26, είδαμε ότι υπάρχουν δύο τροπολογίες σχετικά με την τροποποίηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων ε, για την επανεισαγωγή συνοριακών ελέγχων σε περίπτωση που εντοπιστούν ε, σημαντικές ελλείψεις ε, στο πλαίσιο της περιοχής Σέγγεν. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι η η λήψη των αποφάσεων αυτών με, την, με εφαρμοστικές πράξεις από την Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό θέμα για μας. Ε, ευχαριστώ η, ε, Δανέζικη Προεδρία. Ε, η Προεδρία θα ήθελε και αυτή να ευχαριστήσει την εισηγήτρια καθώς και τους άλλους ευρωβουλευτές που έχουν υποβάλει τροπολογίε. Πιστεύουμε αποτελεί πολύ καλή βάση το σχέδιο έκθεση ε, για την πρόθεση του σημαντικού αυτού θέματο. Οι εργασίε πάνω στην πρόταση ήδη έχουν ολοκληρωθεί. Ε, ε ήδη έχουν προχωρήσει συγγνώμη, στην ομάδα εργασία ε, του Συμβουλίου. Ε, ωστόσο, η ομάδα εργασία δεν είχε τη δυνατότητα να εξετάσει αναλυτικά την, το σχέδιο έκθεση και τι τροπολογίε. Αλλά για μένα είναι προφανέ ότι όσον αφορά την λήψη αποφάσεων για την επανεισαγωγή ε, ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα σε εξαιρετικέ περιστάσει. Ε, η Επιτροπή σα και το Συμβούλιο έχουν ε, την ίδια προσέγγιση, παρόμοια προσέγγιση. Είναι σημαντικό ο έλεγχο των συνόρων για τα κράτη-μέλη και για λόγου ασφαλεία. Από την άλλη, ε, η ελεύθερη κινητικότητα των ανθρώπων ε, είναι μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και θέλουμε να διασφαλίσουμε την διαφάνεια και την καλή διακυβέρνηση. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τις ιδέες τους και προσλέπουμε στον, διάλογο, στον προσεχή διάλογο πάνω στην πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε τώρα ένα κατάλογο βουλευτών. Ο κύριος Κοέγιο καταρχήν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με δύο αρχές. Καταρχήν, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, όχι στο κοινοβούλιο μας, που εξετάζουν το θέμα αυτό, ως τον εύκολο τρόπο να επανεισαχθούν οι έλεγχοι στα σύνορα. Εμείς δεν το βλέπουμε έτσι. Θέλουμε να προστατεύσουμε την ελεύθερη κινητικότητα των πολιτών. Και αυτό είναι ο πρωταρχικό μας στόχο. Αυτό σημαίνει ότι η επανεισαγωγή ελέγχων στα σύνορα θα πρέπει να είναι μέτρο ε, εξαιρετικό, ε, προσωρινό, ε, να αποτελεί την ίστατη λύση και, ως, και να αποτελεί αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένη διαδικασία. Και γι' αυτό οι δύο αυτές εκθέσεις, η δική μου και της κυρίας Βέμπερ, συνδέονται μεταξύ τους, διότι δεν θέλουμε εδώ στο Κοινοβούλιο να να δούμε επανεισαγωγή των ε, συνόρων ε, εκτός της διαδικασίας αξιολόγησης. Η δεύτερη αρχή, ε, την οποία θέλω να θυμίσω στους συναδέλφους, είναι ότι τα σύνορα είναι κοινό θέμα, αλλά εθνική αρμοδιότητα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στις εθνικές, ισορροπίες, στις εθνικές αρμοδιότητες για το ελέγχου στα σύνορα και το κοινό συμφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε είναι το ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του κάθε θεσμικού οργάνου. Να το κάνω πιο σαφές αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στη διαδικασία αξιολόγησης. Γιατί διότι η ε, αξιολόγηση ομοτήμων δεν λειτουργήσε. Ξέρουμε ότι δεν λειτουργήσε διότι τίποτα δεν συνέβη όταν εντοπίστηκαν προβλήματα στα σύνορα. Ε, επί αρκετά χρόνια ε, παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα χωρίς να γίνει τίποτα. Δεν λειτουργήσε λοιπόν η αξιολόγηση ομοτήμων. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία αξιολόγηση ε, με αρμοδιότητε προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με διαφάνεια. Ε, όπου να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο και ελπίζουμε με τη διαδικασία αυτή να βελτιωθούν τα πράγματα όσον αφορά τους ελέγχους στα σύνορα. Το πρόβλημα όμως είναι πάντα το ίδιο. Τι θα κάνουμε Εάν αντιμετωπίσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή στο σύνολο της περιοχής Σέγγεν. Η πρώτη μας ε, προσέγγιση θα πρέπει να είναι παιδαγωγική, να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη μέσω της Frontex, μέσω ευρωπαϊκών οργανισμών, ε, σε κάποιες περιπτώσεις με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση από τα σχετικά ταμεία. Εάν όμως ε, ε, αν παραμείνει το πρόβλημα, θα πρέπει να ε, εξετάσουμε την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μέχρι να λυθεί το θέμα. Ποιο θα λάβει τέτοια απόφαση. Είδα τι διάφορε προτάσει. Και υπάρχουν ε, ουσιαστικά δύο ιδέες στις τροπολογίες. Είτε το Συμβούλιο, να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες το Συμβούλιο, υπάρχουν τροπολογίες που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση, ή η Κομισιόν. Να είμαι ειλικρινής θα τα πω λίγο χοντρά, Εμένα δεν μου αρέσει καμία από τις δύο προτάσεις. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει ούτε με την διαδικασία της επιτροπολογίας. Το είπα αυτό στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, πριν κάποιους μήνες. Δεν νομίζω ότι η διαδικασία της επιτροπολογίας είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Γιατί, διότι δεν είναι διαφανής η διαδικασία αυτή. Ούτε πιστεύω ούτε εάν δοθούν τα εκτελεστικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε αν δοθούν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται για διαδικασίες όπου δεν συμμετέχει στην πραγματικότητα το κοινοβούλιο μας. Αυτό που προτείνω και γι' αυτό έχω υποβάλει σχετική τροπολογία είναι μια πιο διαφανή διαδικασία. Η επαναφορά ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα θα πρέπει να αποτελεί προνόμιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή η πρωτοβουλία θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση με το Κοινοβούλιο και η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται από το Συμβούλιο. διότι η αρμοδιότητα των εξωτερικών συνόρων ε, εξακολουθεί να είναι εθνική αρμοδιότητα και δεν νομίζω ότι θα είναι σοφό, ούτε νομίζω ότι θα είναι δυνατόν να αφαιρέσουμε από το Συμβούλιο αυτή την αρμοδιότητα. Κλείνοντας λοιπόν κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό προφίλ της διαδικασίας αυτής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανισμοί, όπως προβλέπεται σε αρκετές τροπολογίες, θα πρέπει να παίζουν πιο αποτελεσματικό ρόλο, όμως Εάν ως ίστατη λύση πρέπει να επαναφέρουμε τους ε, ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα. Η διαδικασία θα πρέπει να είναι πρωτοβουλία της Κομισιόν, ε, συμβουλευτικός ρόλο του Κοινοβουλίου και τελική ε, οριστική απόφαση με ειδική πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σένσιου. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την συνάδελφό μας την κυρία Ρενάτε Βέμπερ για τον τρόπο ε, σύνταξης της έκθεσης αυτής και τον ε, τρόπο ε, που χειρίζεται τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα θεσμικά όργανα στις τελικές φάσεις διαπραγμάτευση πάνω στην έκθεση αυτή. Θα ήθελα επίσης να την ευχαριστήσω για τον τρόπο που καταφέραμε να συνεργαστούμε μέχρι τώρα και που νομίζω θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, Συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος Κάρλος μέχρι τώρα. Όχι κατά 100% αλλά σε μεγάλο βαθμό συμφωνώ με αυτά που είπε. Θα συζητήσουμε, θα εξετάσουμε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να προτείνουμε συμβαστικές τροπολογίες που να είναι αποδεκτές από όλους. Ε, τις τροπολογίες εγώ θα τις χώριζα σε τρεις κατηγορίες. Καταρχήν έχουμε κάποιες τροπολογίες οι οποίες διασαφηνίζουν κάποιες διατάξεις στην πρόταση της Επιτροπής. Έχουμε αυτή που αναφέρεται στις κατευθυντήρες γραμμές και την ετήσια έκθεση που θα πρέπει να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο. Η έκθεση αυτή, κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τι δραστηριότητε που συνδέονται με την περιοχή Σέγγεν. Η δεύτερη κατηγορία τροπολογιών που είναι σημαντική για την πολιτική μου ομάδα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι σημαντική και για τις άλλες πολιτικές ομάδες είναι οι τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την ε, εξάλληψη οποιαδήποτε σύγχυση όσον αφορά την ε, μεταναστευτική ροή ως πιθανό λόγο για την επαναφορά συνοριακών ελέγχων. Η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την επαναφορά ελέγχων στα σύνορα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ευρωπαϊκά μέσα τα οποία να μας επιτρέπουν διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Η διαχείριση των ροών αυτών θα πρέπει να γίνεται με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ε, θα πρέπει όμως ε, οι μεταναστευτικές ζωές αποτελούν δικαιολογία για τον περιορισμό ε, της ελεύθερης κινητικότητας στην περιοχή Σένιαν. Και η τελευταία κατηγορία τροπολογιών, όπως είπε και ο συνάδελφος Κάρλος, είναι ασχολούνται με τις περιπτώσεις όπου θεωρείται απαραίτητη η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μετά τον εντοπισμό σημαντικών ελλείψεων στο μηχανισμό Σέγγεν. Προτείνουμε σε περίπτωση που τα συμπληρωματικά μέτρα δεν ήταν αποτελεσματικά η Επιτροπή να ε, διαβιβάζει έκθεση στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, όπου θα επιβεβαιώνει την ανάγκη για την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα έχουν ένα μήνα για να ε, εκδώσουν ομοδότηση για, πάνω στην έκθεση αυτή και κατόπιν η Κομισιόν θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει σχετικά με την προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα σύνορα με εκτελεστική πράξη σύμφωνα με την ε, διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό, αυτή θα είναι η κατάλληλη λύση. Θα ε, συνομιλήσω με τον συνάδελφο Κάρλος για να δούμε ποια από τις δύο προτινόμενες λύσεις είναι καλύτερη. Όπως και να έχει, ο μηχανισμός που προτείνω επιτρέπει ε, δημοκρατικό έλεγχο, αποτελεσματικό δημοκρατικό έλεγχο της διαδικασίας και σε κάποιες ακραίες, σε ακραίες, στις ακραίες περιπτώσεις όπου θα είναι απαραίτητη η προσωρινή επαναφορά των ελέγχων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την Σκιώδη σήμερα που δεν μπορεί να παραβρεθεί. Συνολικά εμείς οι πράσινοι πιστεύουμε ότι το Σέγγεν ε, θα είναι ένα κοινοτικό μέσο και θα πρέπει ρήποτε δυνατότητα επαναφορά των ελέγχων να ε, μπορεί να γίνει σε επίπεδο κοινοτικό. Κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έχει ποτέ συμβεί. Δεν ναι, βλέπω λοιπόν τη βελτίωση προσφέρεται εδώ. Συμφωνούμε λοιπόν ότι οι μεταναστευτικές πιέσεις ε, δεν αποτελούν απειλή στα εξωτερικά μας σύνορα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να φέρονται ως αιτία, ως λόγος για την επαναφορά των ελέγχων. Ε, θα καταθέσουμε μια τροπολογία σχετικά με την ενημέρωση του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο άμεσα θα πρέπει να ενημερώνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. Πιστεύουμε ότι η Κομισιόν είναι πολύ ασαφής στο να αναφέρει πότε υπάρχει απειλή στην εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει πάντα μια απειλή όπως η τρομοκρατία κλπ. Αλλά χρειάζεται να υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο, το απτό σε ό,τι φορά την λόγο απειλή. Και αυτό θα πρέπει να φυσικά να αποδεικνύεται. Η Κομισιόν προτείνει πως αποτυχίες στην ε, πολιτική επιστροφών θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναφορά των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα και κρίνουμε ότι αυτό δεν είναι σωστό γιατί, γιατί πέραν των ελλείψεων που υπάρχουν στην πολιτική επιστροφών Θεωρώ ότι θα πρέπει να δούμε και τα άτομα τα οποία εμπλέκονται σε αυτές τις πολιτικές επιστροφών. Ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα όπου το κοινοτικό επίπεδο θα είναι αυτό το οποίο θα εμπλέκεται όταν χρειαστεί να ληφθεί απόψη και να μην θεωρήσουμε ότι οι μετανάστες αποτελούν απειλή στην εσωτερική ασφάλεια των χωρών μας. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ένστε, ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο το θέμα. Πραγματικά, φυσικά, επικροτούμε ε, το Σέγγεν ε, πέρα από τα προβλήματα που ε, αντιμετωπίζουμε, διότι η ελεύθερη κινητικότητα είναι τόσο σημαντικό αγαθό ε, και σύμβολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι πολύ δύσκολο να το αγγίξουμε. Στην περίπτωση αυτή όμως νομίζω ότι το περιθώριο ε, διακριτικής ευκαιρίας των κρατών μελών να είναι όσο γίνεται πιο στενό. Ε, εγώ πιστεύω ότι το μόνο λογικό είναι η κοινοτική μέθοδος ε, για να αποφύγουμε την αυθαιρεσία. Στην, στο άρθρο 23 του κώδικα Schengen υπάρχουν ε, συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Και πιστεύουμε ότι αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν ε, προς την κατεύθυνση της κοινοτικής μεθόδου. Της κοινοτικής μεθόδου. Ε, καταλαβαίνουμε κυρία Βέμπερ τι δυσκολίες ε, έχετε. Ε, έχουν υποβληθεί και πολλές τροπολογίες. Εάν κάτι θέλουμε να αλλάξουμε, να αλλάξουμε προς την κατεύθυνση της κοινοτικής μεθόδου και να κοιτάξουμε εάν ε, έχουμε τις σωστές προτάσεις μπροστά μας. Αν συμφωνήσουμε να ακολουθήσουμε την κατεύθυνση αυτή, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ε, ξανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Ναι, η πρωτοβουλία θα πρέπει να είναι της Κομισιόν, ναι, συμφωνώ απόλυτα, όχι του Συμβουλίου. Γενικά πιστεύουμε ότι ο έλεγχος στα σύνορα θα πρέπει να επανεισάγεται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, ε, σε περίπτωση, τι να σας πω, ε, εξοκοσμικού κινδύνου. Ε, σε μια από τις ε, τροπολογίες μας, όπως και η πράσινη, μιλάμε για ε, σοβαρή και συγκεκριμένη απειλή. Θα πρέπει να καθορίζεται επίσης ο ρόλος του κινδύνου αυτού. Καταλαβαίνουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η συγγήτρια να λάβει επαρκώς υπόψη της την πτυχή της μετανάστευσης. Έχουμε την ε, τροπολογία 5. Αναφέρονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών ε, και η ε, δημόσια ασφάλεια, αλλά δεν νομίζω ότι έχει βαθύνει επαρκώς το θέμα. Οι άλλες τροπολογίες είναι πολύ αυστηρές όσον αφορά τον μηχανισμό επιστροφής. Εάν υπάρχουν ελλείψεις στις επιστροφές, αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θα πρέπει να ε, συνδέσουμε μεταξύ τους τα δύο αυτά θέματα. Και τέλος, υπάρχουν και κάποιες ε, μικρές τροπολογίες που έχουν ε, να κάνουν με την ενημέρωση του κοινού στην περίπτωση της επαναφοράς των ελέγχων. Γενικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το, ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και όπως σας είπα οτιδήποτε ακολουθεί την κοινοτική μέθοδο οτιδήποτε αποτρέπει τα κράτη-μέλη από το να, ε, να κινούνται μόνα τους ε, μας βρίσκει σύμφωνος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σταπκόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βέμπερ για τη δουλειά που έχει επιτελέσει. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της επαναφοράς των ελέγχων. Η Πολωνία είναι μία από τις χώρες που εισήλθε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρισκόμαστε και εμείς, έχουμε ενταχθεί δηλαδή στον Σέγγεν, χώρο Σέγγεν και αυτό για τους Πολωνούς πολίτες αποτελεί ένα μεγάλη ικανοποίηση, μεγάλο προνόμιο που μπορούν, να διασχίζουν τα σύνορα ελεύθερα. Εάν λοιπόν επαναφέρουμε τα, τους ελέγχους, αυτό θα γίνει αισθητό με τρόπο όχι ιδιαίτερα Θα ήθελα να ζητήσω την τελική απόφαση να την λάβει το Συμβούλιο. Η Κομισιόν μπορεί να κάνει σχετική ανάλυση, αλλά η τελική απόφαση θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια του Συμβουλίου. Αυτό περιλαμβάνεται και σε μια τροπολογία που έχω καταθέσει. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο δεν μας απασχολεί σήμερα, αλλά την προσεχή εβδομάδα θα ζητήσουμε από την Κομισιόν να εξετάσει όλα αυτά τα στοιχεία και ειδικά να εξετάσει το ζήτημα των κοινών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Ε, αναφέρομαι σε περιπτώσεις ε, τις οποίες υπάρχει ένας πολίτης ο οποίος ε, ζει δίπλα στα σύνορα με την Ουκρανία, αλλά θα πρέπει να έχουμε λοιπόν ένα πιο απλουστευμένο σύστημα διέλευση των σύνορων. Κυρία Μάκεντάιρ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχήν την κυρία Βέμπερ θερμά για την εργασία της και στηρίζω την προσπάθειά της. Η σημασία της ελεύθερης κυκλοφορίας, κάτι το οποίο όλοι υποστηρίζουμε, Χρειάζεται όμως να βρεθεί κάποια ισορροπία, να υπάρχουν δηλαδή κάποιες δυνατότητες, να προσφέρουν κάποιες δυνατότητες στα κρατη Ως Βρετανή Ευρωβουλευτής κατανοώ τις ευαισθησίες που υπάρχουν σε ό,τι φορά τους ελέγχους στα σύνορα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ξέρετε, έχει διατηρήσει τους ελέγχους αυτούς. Αλλά πολλές αντιπροσωπείες στην ομάδα μου ε, εκφράζουν ανησυχίες και σημείωσαν ανησυχίες ε, της πρότασης αυτής της Κομισιόν. Τρεις τροπολογίες έχουμε καταθέσει και αφορούν ε, στα εκτιμώντας, ε, όχι στο διατακτικό του εγγράφου. Δεν νομίζω όμως ε, ότι υπάρχει, δημιουργούν πρόβλημα. Τροπολογία μου υπαριθμών 33 αναφέρει να λαμβάνουν υπόψη αιτήματα ε, των κρατών μελών για άμεση δράση. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε να γίνουν συνεδριάσεις επί των συνεδριάσεων. Μερικές φορές χρειάζεται να δράσουμε άμεσα. Αυτή η τροπολογία λοιπόν θα μας επιτρέψει να τηρήσουμε την ε, απαραίτητη ισορροπία. Ευχαριστώ. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους ε, που εξέφρασαν τις απόψεις τους ε, και μας παρουσίασαν τα επιχειρηματά τους σχετικά με τις τροπολογίες που κατέθεσαν. Ευχαριστώ και την Κομισιόν και το Συμβούλιο για τα παρεμβάσεις τους. Δεν Ήθελα να ξεκινήσω συζήτηση με αναφερόμενη στα όσα έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν, διότι κρίνω πως δεν είναι απαραίτητο τώρα, τώρα πια. Βρισκόμαστε σε μια διαφορετική φάση. Αλλά ίσως θα ήταν ορθό να υπενθυμίσω στους συναδέλφους πως όσο και αν εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση της Κομισιόν, διότι ε, συμφωνεί με την ε, κοινωνική προσέγγιση του Σέγγεν καταλαβαίνετε ότι μερικές φορές είναι καλύτερο να σκέφτεται κανείς με το μυαλό και όχι με την καρδιά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να δεχτούν οι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, αλλά δεν θα δεχθεί το Συμβούλιο. Πρέπει λοιπόν να ε, βρούμε κάτι το πιο εφικτό θα λέγαμε, προκειμένου να γίνει δεκτό. Και αυτό θα είναι σίγουρα καλύτερο αυτό που έχουμε τώρα. Μιλάμε για ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή και ειλικρινά άμα κοιτάξουμε γύρω μας και δούμε πόσο οι πολίτες θέλουν να διατηρηθεί το Σέγγεν τους ικανοποιεί οι τελευταίες δηλώσεις για τις εξελίξεις στην ζώνη Σέγγεν δεν ε, ήταν ε, οι κατάλληλες. Ε, κοιτάξτε, τα μεταναστευτικά ρεύματα δεν πρόκειται να θεωρηθούν ως απειλή στην εθνική ασφάλεια. Αυτό το ανέφερα ευθύς εξ αρχής, αναφέρεται και στο έγγραφό μου, καθώς και επίσης και η διαδικασία επιστροφών δεν θα πρέπει να σχετίζεται με την δημόσια, με την ε, δημόσια ασφάλεια ή την απειλή στη μια χώρα. Άρθρα 24-25, τροπολογίες σχετικές, ε, τροπολογίες και στα εκτιμώντας, παραμένει όμως το ζήτημα του 26 εδώ είτε θα πρέπει να υπάρξει η επιτροπολογία είτε μιας άλλη μορφής απόφαση. Και αυτό σίγουρα θα γίνει αντικείμενο περαιτέρω συζητήσεων με τους σκιώδεις, με το Συμβούλιο, με την Κομισιόν και προγραμματίζω φυσικά να οργανώσω το σύντομο των δυνατών μια συνεδρίαση με τους σκιώδεις ηγητές ώστε να καταρτήσουμε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και να διασφαλίσουμε πώς τα πράγματα θα εκτεληχθούν προς την σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Από εδώ και στο εξή θα παραμείνουμε σε επαφή, αλλά και μετά από τις ψηφοφορίες διότι πρέπει να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ για τη δουλειά που κάνατε και την εργασία που πρόκειται να κάνετε στο εγγύς μέλλον. Θα αναζητήσετε συμβαστικές τροπολογίες οι οποίες συμβαστικές τροπολογίες θα μας επιτρέψουν να προγραμματίσουμε την ψήφιση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τον Απρίλιο. Ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 18 και 19. Ομού κοινή συζήτηση. Σημείο 18. Αυτό αφορά την πρόγραμμα δράση του νομίου ανταλλαγών, τη συνδρομή και τη κατάρτιση για την προστασία του ευρώ από την παραχάρευση και την κυβδηλία πρόγραμμα Πέρικλεις ε, 2020. Εδώ η συγγήτρια είναι η κυρία Άνθια Μάκεντάερ. Και επίσης θα συζητήσουμε το σημείο 19 για την επέκταξη του κανονισμού για τη θέσπιση προγράμματος δράσης σε θέματα κατάρτισης, ανταλλαγών και συνδρομής για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη πρόγραμμα Περικλής σε ό,τι αφορά φυσικά τα κράτη-μέλη που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ ως ενίο νόμισμα. Εδώ εισηγητή έχουμε τον κύριο Αγκουστίν Δίας Δεμέρα, ο οποίος όμως απουσιάζει και θα τον αντικαταστήσει ο κύριος Κάρλος Κοέλιο. Λοιπόν, ας ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και μια ανταλλαγή απόψεων το λόγο έχει η Κομισιόν. Ο κύριος Χόου νομίζω, αν προφέρω σωστά. Χάου. Χόου. Από την Όλαφ ε, θα μας παρουσιάσει την πρόταση και θα ακούσουμε την Δανική Προεδρία του Συμβουλίου. Θα ακούσουμε την κυρία μάκεντάρ και τον κύριο Καλοσκολιά και θα ακολουθεί συζήτηση. Κύριε Χάου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι εξαιρετική αυτή η ευκαιρία για την Επιτροπή να παρουσιάσει την πρότασή της Περικλής 2020 ε, για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κυβδηλία. Ε, ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος αυτού, όπως σας είπα, είναι ένα ε, πρόγραμμα κατάρτισης, ανταλλαγής προσωπικού, ε, δικτύωσης, ευαισθητοποίησης για να βελτιωθεί η προστασία του ευρώ από την παραχάραξη. Έχουμε ειδικέ ομάδες επιλέξιμων δικαιούχων, ε, τις, εθνικές, τις αρμόδιες εθνικές αρχές για ε, την καταπολέμηση της κυβδηλίας ε, του ευρώ. Επίσης εκπροσώπους ε, των εθνικών τραπεζών, των νομισματοκοπίων και από επιστημονικά εργαστήρια τα οποία είναι σε θέση να εντοπίζουν τα παραχαραγμένα χαρτονομίσματα και νομίσματα. Έχουμε λοιπόν ε, επαγγελματικό υπόβαθρο για την καταπολέμηση της κυβδηλίας. Γιατί το πρόγραμμα Περικλής 2020 χρειαζόμαστε συνέχιση της ε, υποστήριξης και προστασίας του ευρώ εντός αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απειλή κυβδηλίας παραμένει υψηλή. Το ευρώ έχει διεθνή διάσταση ως νόμισμα δεδομένης αυτής της ε, διεθνούς διάστασης είναι απαραίτητο ε, να καταπολεμήσουμε τις επαγγελματικές οργανώσεις ε, σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε λοιπόν να εξελίσσουμε τα τεχνικά μέσα για την καταπολέμηση της κυβδηλίας, συμπληρώνοντας τις προσπάθειες που καταβάλουν τα κράτη-μέλη. Επίσης έχουμε εντοπίσει ε, κάποιες ε, απειλές που τώρα εμφανίζονται στον κόσμο εκτός της Ευρώπης, ε, στην Κίνα για παράδειγμα. Η δράση σε επίπεδο ευρωπαϊκό είναι συμπληρωματική σε σχέση με αυτά που ήδη κάνουν τα κράτη-μέλη. Έτσι διασφαλίζεται ομοιογένεια κατά την προστασία του ευρώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ο λόγος που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει δύο προτάσεις. Η μία καλύπτει με τις προτάσεις της ε, τα κράτη-μέλη που έχουν εισάγει το ευρώ, το κοινωνόμισμα. Και έχουμε και μία πρόταση που καλύπτει τα κράτη-μέλη που δεν έχουν εισάγει ακόμα το ευρώ ως ενιαίο νόμισμα. Το σχέδιο κανονισμού καθορίζει σαφείς στόχους. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο βασικός στόχος είναι η προστασία του ευρώ, των νομισμάτων και χαρτονομισμάτων του ευρώ από την κυβδηλία και την παραχάραξη. Πόσο, πώς το κάνουμε αυτό, επαναλαμβάνομαι, αλλά με ανταλλαγή πληροφοριών, με κατάρτιση, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ε, και με επιστημονική και αναλυτική δουλειά για την βελτίωση μεθόδων εντοπισμού παραχαραγμένων νομισμάτων. Έχουμε αρκετά σημαντική ιστορία. Υπήρξε πρόγραμμα Περικλής 1 και Περικλής 2. Το αρχικό πρόγραμμα δημιουργήθηκε με απόφαση του Συμβουλίου του 2001. Η απόφαση αυτή ε, τροποποιήθηκε ώστε να παραταθεί ε, για το διάστημα των δημοσιονομικών πρακτικών 2007-2013. Έχουμε πετύχει αυτά αποτελέσματα, 84 δράσεις είχαμε, 93% του προϋπολογισμού έχει διατεθεί 4.000 ε, συμμετέχοντες είχαμε. Και σύμφωνα με ε, τις ανταποκρίσεις που, που λάβαμε, το 98% των ε, συμμετεχόντων ήταν ε, αρκετά ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα. Συζητάμε σε τακτική βάση, σε τήσια βάση με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Europol, την Interpol. Ε, συζητάμε λοιπόν μαζί τους ε, το ετήσιο ε, πρόγραμμα εργασίας ε, του Περικλής. Συζητάμε τη στρατηγική αυτή με τα κράτη-μέλη και τα άλλα θεσμικά, και τα άλλα θεσμικά όργανα ε, στα πλαίσια των εργασιών για την παραχάραξη του ευρώ. Η έμφαση φυσικά θα πρέπει να δίδεται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε όμως μια συγκεκριμένη προτεραιότητα για την ε, ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας. Ε, καταφέραμε στην νότιο-ανατολική Ευρώπη να ε, δημιουργήσουμε μια τέτοια συνεργασία για να στοχεύσουμε σε χώρες που εποφελούνται ή που παράγουν μεγάλο αριθμό παραχαραγμένων νομισμάτων. Με αυτήν την ε, πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ε, λοιπόν δημιουργούμε τώρα ε, ανάλογη πλατφόρμα για την Βόρειο-Δυτική Ευρώπη. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής μας του ευρώ. Έχουμε και ε, δικτύωση εκτός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Έχουμε επαφές ε, με την Ειδική Υπηρεσία κατά της παραχάραξης ε, στη Μαδρίτη για να καλύψουμε και τη Λατινική Αμερική. Γιατί? Διότι έχουμε διαπιστώσει τουλάχιστον ότι παράδειγμα, για παράδειγμα στην Κολομβία ε, παράγεται σημαντικός όγκος παραχαραγμένων νομισμάτων και ευρώ και δολαρίων. Ε, αυτό συνδέεται με ε, το ε, εκτενές οργανωμένο έγκλημα στη χώρα αυτή που και τις δραστηριότητες νομοποίησης παράνομων εσόδων και άλλων εγκλημάτων. Επίσης θέλουμε να εξετάσουμε και τι γίνεται στη Ρωσία όσον αφορά τη νέα πρόταση του 2020, για το 2020. Προτείνουμε τώρα έναν κανονισμό με ένα οριζόντιο μέρος σε μια βασική πράξη σύμφωνα με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ε, έτσι θέλουμε να βελτιώσουμε την ε, νομική βεβαιότητα. Έχουμε απλοποιήσει την πρόταση. Έχουμε εισάγει επίσης ε, τις διατάξεις ε, για τα, τις επιλέξιμες δαπάνες. Ένα δεύτερο θέμα πιο ουσιαστικό είναι ότι έχουμε αυξήσει το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 90% σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επιτρέποντα έτσι στο περιφερειακό στοιχείο στο οποίο μόλις ανέφερα, όταν μιλάμε για την πλατφόρμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ουσιαστικά καλούμε τα κράτη-μέλη να παρουσιάσουν προτάσεις. προσπαθώντας έτσι να ε, τα κινητοποιήσουμε. Γνωρίζουμε τις, ε, τους δημοσιονομικούς ε, περιορισμούς πολλών χωρών στην περιοχή αυτή. Γι' αυτό αυξήσαμε το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 90% σε κάποιες περιπτώσεις με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος σχετίστηκε και το ότι τώρα προτείνουμε ε, συμφωνίες για την αγορά εξοπλισμού. Ε, κάτι που πρέπει να συνδυαστεί με ε, συντήρηση του εξοπλισμού και με ανάλογη κατάρτιση. Είχαμε μία έρευνα των ενδιαφερόμενων ομάδων. Ε, ε, τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής έχουν ε, δημοσιευτεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε την Δανέζικη Επιτροπή επίσης να κάνει μια σύντομη εισαγωγή, προτού να ακούσουμε τους εισηγητές μας. Να πω μερικά λόγια σχετικά με τις δύο προτάσεις περικλής. Στο Συμβούλιο είχαμε δύο συναντήσεις Η πρώτη ήταν παρουσίαση από την Κομισιόν και μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων ε, στα τέλη Φεβρουαρίου και σήμερα το πρωί στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου οριστικοποίησαμε την ε, τεχνική εξέταση των άρθρων και των εκτιμώντας και στόχος της Δανικής Προεδρίας είναι να λάβει μια διαπραγματευτική εντολή μέχρι το τέλος της ε, Προεδρίας μας προκειμένου να ξεκινήσουν τις συζητήσεις με το Ευρωκοινοβούλιο το αυστημότερο και προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο επί του φακέλου αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα σας ακούσουμε τους συζητητές. Η κυρία Μάκεν Τάερ την πρώτη έκθεση. Um, thank you, Mr. Chairman. Um, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερος ευγνώμων uh, στους συναδέλφους που μου έδωσαν ε, την ε, έκθεση αυτή. Είναι η πρώτη φορά που συντάσσω έκθεση. Θα προσπαθήσω να κάνω ώστε να τον καλύτερη δουλειά. Νομίζω ότι ουσιαστικά θα συνεργαστούμε, γιατί εγώ έχω αυτό το ρόλο εδώ, να συντάξω την έκθεση. Και υπάρχει και ο συνάδελφος Ντίαφ ε, μέρα ή τέλος πάντων ο συνάδελφος που τον εκπροσωπεί σήμερα. Θα συνεργαστούμε λοιπόν οι δυο μας. Αν κατάλαβα καλά, το πρόγραμμα Περικλής ήταν ε, το αποτέλεσμα της ε, απόφασης του Συμβουλίου ουσιαστικά και από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης αρχικώς πλέον συμπεριλαμβάνει όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αυτή λοιπόν η επέκταση ε, του πεδίου εφαρμογής προγράμματος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, εξού και υπάρχουν δύο εκθέσει. Τέλο πάντων, αν ε, ζητεί το γνώμη μου, θα έλεγα ότι πιο απλό είναι να έχουμε μόνο μία έκθεση, αλλά τέλος πάντων, αφού έχουμε αυτή τη νομική βάση, πρέπει να έχουμε δύο εκθέσει. Προέρχομαι από το Ενωμένο Βασίλειο. Εμεί δεν είμαστε στο Ενωμένο Βασίλειο μέλη τη ε, ωστόσο, θέλω να καταστήσω σαφέ ότι έχει τεράστια σημασία για το Ηνωμένο Βασίλειο το όλο θέμα. Μπορεί να μην είμαστε στο ευρώ, αλλά ευρώ χρησιμοποιούμε. Ευρύτερα χρησιμοποιείται το ευρώ, επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προσβλέπω στη συνεργασία και με τους υπόλοιπους συναδέλφους για την εκπόνηση της έκθεσης. Είμαι ευγνώμων στον κύριο Χάου από την Όλαφ που μας εξήγησε ιδίως τα καινούργια στοιχεία. Νομίζω ότι όλοι είμαστε υπέρ της απλούστευσης και της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας. Είναι και οι δύο αξιέπαινοι στόχοι. Καλό ήταν επίσης αυτό που ακούσαμε το τελευταίο νέο αποστόματο Συμβουλίου. Οι τελευταίες ειδήσει. Και επαναλαμβάνω προσβλέπω σε απόψεων συναδέλφων και στην καλή μας συνεργασία. Ευχαριστώ. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τώρα και τον κύριο Κοέλιο για τη δεύτερη έκθεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Ντίαθ ε, Ντεμέρα είναι στην Ουάσιγκτον, γι' αυτό και δεν είναι μαζί μας σήμερα. Μου ζήτησε λοιπόν να τον εκπροσωπήσω, κάτι που κάνω ευχαρίστως. Πρώτα απ' όλα θέλω <clears throat> να καλωσορίσω την ε, συνάδελφο Τάιερ και σίγουρα θα συνεργαστούμε Όπως είπε και η κυρία Μακιντάιρ, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες οι δύο εκθέσεις. Δεν μπορεί να στέκει μία χωρίς την άλλη. Καλωσορίζουμε την, την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την επανεξέταση και βελτίωση των μέτρων του προγράμματος Περικλής. Συμφωνούμε και με την επέκταση σε άλλα κρατημέλη και γενικότερα σε όλους τους ε, τομείς. Είναι κάτι θετικό. Αστυνομία, εθνικό νόμισμα, δικαστές, όλα αυτά θα εξασφαλίσουν νομίζω την μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία του ευρώ από κύβδηλα και παραχαραγμένα νομίσματα. Ο κύριος Δίας Δεμέρα λέει ότι ξεκάθαρα έχουμε δει την επιτυχία του προγράμματος Περικλής. Γιατί το ευρώ είναι το λιγότερο παραχαραγμένο νόμισμα στον κόσμο. Σίγουρα υπάρχουν νέες προκλήσεις, υπάρχουν νέες απειλές. Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, ίσως και η ένταξη μελλοντική και άλλων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας υποχρεώνει να προσαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα. Ο κύριος λοιπόν Δίας Δεμέρα καλωσορίζει τις προτάσεις ε, που έχουν γίνει και οι οποίες αναμφίβολα θα έχουν ως αποτέλεσμα την ε, βελτίωση της δράσης και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των ε, υπηρεσιών αντιμετώπισης παραχάραξης. Ευχαριστώ. Contribute. Κύριε Παπαδοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, είμαι σκιώδη εισηγήτρια για, για λογαριασμό τη Προοδευτική Συμμαχία Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Θεωρώ ότι και οι δύο κανονισμοί είναι πολύ σημαντικοί, γιατί ακριβώ θα καταπολεμήσουν την κυβδηλία και την παραχάραξη του ευρώ τόσο στι χώρε ε, στι οποίε χρησιμοποιείται ω νόμισμα, αλλά και σε άλλε χώρε που πιθανόν να ενταχθούν στο μέλλον στην Ευρωζώνη. Ε, από κάποια στοιχεία που έχω δει φαίνεται ότι υπάρχει παραχάραξη ε, κυρίως σε τραπεζογραμμάτια και μάλιστα εκείνα τα τραπεζογραμμάτια που είναι χαμηλής νομισματικής αξίας των 20 ευρώ γιατί ε, αυτά χρησιμοποιούνται πιο πολύ και πλατιά από τους πολίτες. Και είναι σημαντικό ακριβώς να υπάρχουν οι μηχανισμοί. Η εμπειρία από το πρόγραμμα Περικλής από το 2001 μέχρι σήμερα ήταν πολύτιμη Υπάρχουν όντως οι μηχανισμοί και επαγγελματική κατάρτιση και θεωρώ εφόσον το ευρώ εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστικό στόχο των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες ε, χώρε, επιβάλλεται ο συντονισμό σε υπερεθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση τη παραχαράξη. Ε, ο Επίτροπο Σεμέτα, που είναι και αρμόδιο για το θέμα, έχει πει ότι η απάτη σε βάρος του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί έγκλημα χωρίς θύματα. Και όντως ε, αυτή η παραχάραξη ε, σημαίνει ότι τα χρήματα όλων μας, των Ευρωπαίων πολιτών, κινδυνεύουν. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στο μέσο μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, πρέπει να προστατεύσει τα έσοδά της, να βεβαιωθούμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εποφελούνται όσο το δυνατόν περισσότερων από τα κοινοτικά ταμεία μέσα από το πρόγραμμα Περικλής 2020 ε, θα αναδειχθεί για μια ακόμη φορά η ευρωπαϊκή διάσταση της προστασίας του ενιού, του νομίσματος και βέβαια ε, αυτό δεν φύγει ε, τις αρμοδιότητες των κρατών μελών ε, γιατί ακριβώς ακολουθείται η αρχή της αναλογικότητας. Το άρθρο 13 της πρότασης έχει βαρύνουσα σημασία γιατί γίνεται λόγος για προληπτικά μέτρα κατά τη απάντηση τη διαφθορά και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, με τη διενέργεια αποτελεσματικών ελέγχων αλλά και με την επιβολή κυρώσεων. Και αυτέ οι κυρώσει πρέπει να γίνονται. Επίση, ε, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η διευκόλυνση τη πρόσβαση των αρμόδιων εθνικών αρχών των κρατών μελών στο πρόγραμμα και την εφαρμογή σε τρίτε χώρε και να υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μέσω του προγράμματο Περικλή 2020. Θέλω να επισημάνω επίση σε κατακλείδαν το εξή. Η συνεχή εκπαίδευση του ειδικευμένου προσωπικού για την παραχάραξη και την κυβδηλία του ευρώ είναι πολύ σημαντική. Εξίσου σημαντική όμω είναι και η διαρκή ενημέρωση των απλών πολιτών. Και εδώ ακριβώ ήθελα να θέσω μια ερώτηση στον εκπρόσωπο τη Κομισιόν, εάν στη χρηματοδότηση του προγράμματο προβλέπονται και εκστρατείε ενημέρωση του απλού κόσμου σχετικά με την παραχάραξη και την κυβδηλία του ευρώ. Γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν και να προστατεύονται. Okay. Any other members? Willing... Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελα να λάβει μέρος σε αυτή τη συζήτηση. Δεν βλέπω να σηκώνονται χέρια. Δεν νομίζω ότι θέλει κάποιος το λόγο. Άρα, αν θέλουν να προσθέσουν οι συγγητές μας κάτι, μπορώ να τους δώσω το λόγο ή όχι. Να σταματήσουμε εδώ προς το παρόν. Ωραία. Αυτό ήταν λοιπόν η πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εισηγητών, σκιωδών εισηγητών. Ακούσαμε την ε, απόψη της σκιώδου εισηγητρίας κυρίας Παπαδοπούλου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση και για μία φορά εκτάκτος είμαστε πολύ μπροστά στο χρονοδιάγραμμα. Έχουμε το σημείο 20 για τις ποινικέ κυρώσεις, για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, για το οποίο υποτίθεται ότι θα έχουμε παρουσίαση της Επιτροπής. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής όμως δεν έχει φτάσει ακόμη. Για μια ακόμη φορά λοιπόν θα πρέπει να διακόψουμε, αυτή τη φορά για μισή ώρα. Λυπούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για όσους ε, έχουμε επιβιώσει αυτές τις δύο ημέρες ε, συνεδριάσεων. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα και εγώ λυπάμαι, αλλά τι να κάνω. Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προγραμματιστεί να είναι εδώ στις 6 για αυτό το θέμα, 6 το απόγευμα έτσι, θα πρέπει να του περιμένουμε για μισή ώρα, αν θέλουμε να ακούσουμε την παρουσίαση του θέματος που θα είναι και το τελευταίο της απόψινης συνεδρίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Yes, Τελευταίο θέμα της μακράς αυτής ημέρας. Να συζητήσουμε τις ποινικέ κυρώσει για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικέ πληροφορίε και τις πράξεις χειραγώγησης τη αγοράς. Ας ακούσουμε την παρουσίαση της Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει ένα πακέτο μέτρων σε μια πρόταση οδηγία για τι ποινικέ κυρώσει για τι πράξει προσώπων που κατέχουν αντιπιστευτικέ πληροφορίε και τι πράξει χειραγωγήσει τη αγορά. Αυτή είναι η παρουσίαση που θα ακούσουμε. Α ακούσουμε λοιπόν την Κομισιόν και κατόπιν θα έχουμε συζήτηση. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα, που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε αυτή την ε, πρόταση. Θα είμαι πολύ σύντομη. Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε στο τέλος της ε, δεύτερης ημέρας συνεδρίασης της ΛΥΜΠΕ. Θα το λάβω αυτό υπόψη μου λοιπόν κατά διάρκεια της ε, παρουσίασής μου. Ε, κατά τη γνώμη μας η πρόταση αυτή είναι πολύ επίκαιρη, διότι δύο χρόνια έχουν περάσει από την ε, θέση σε ισχύ της συνθήκη τη Λισαβόνα και αρχίζουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα ε, της εργασίας αυτής. Και η πρόταση αυτή αποτελεί μέρος της πολιτικής μας για το ποινικό δίκαιο και μάλιστα είχε ανακοινωθεί στην ανακοίνωσή μας για το ποινικό δίκαιο που, είχε, που είχαν παρουσιάσει στην Επιτροπή σας. Για πρώτη φορά λοιπόν εφαρμόζουμε τις ε, αρχές ε, για να διασφαλίσουμε την ε, συνεπή αντιμετώπιση των πράξεων προσώπων που κατέχουν επιστημονικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγωγής αγοράς. Πρώτη φορά χρησιμοποιείται η συνθήκη για να προταθούν κυρώσεις για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών σύμφωνα με το ε, άρθρο 83.2. Η πρότασή μας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου που περιλαμβάνει μια, έναν μητρικό κανονισμό, να το πούμε έτσι, για την ε, χειραγώγηση της αγοράς ε, και τώρα έχουμε την συνοδευτική πρόταση με τις ποινικέ κυρώσεις που στόχο έχει να ενισχύσει τους ουσιαστικούς κανόνες κατά την, της χειραγώγησης της αγοράς καθώς και το καθεστώς διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Με βάση την ε, μελέτη αντικτύπου μας, ε, στόχο ε, είχαμε να ασχοληθούμε με την χειραγώγηση της αγοράς σε ένα μέσο που έχει να κάνει με τις ποινικέ κυρώσεις. Στην ανακοίνωσή μας για το ποινικό δίκαιο έχουμε παρουσιάσει τις αρχές τις οποίες ακολουθούμε. Οι ποινικές κυρώσεις αποτελούν ίστατο μέτρο. Τα ε, ποινικά μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να είναι ουσιαστικά σύμφωνα με το άρθρο 83 και βέβαια ε, η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει να γίνεται σεβαστή καθότι ενεργούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί λοιπόν προτείνουμε ευρωπαϊκούς κανόνες, ευρωπαϊκές κυρώσεις για να αντιμετωπίσουμε τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγωγής αγοράς. Το θέμα είναι η ακεραιότητα της αγοράς και η εμπιστοσύνη του κόσμου στις αγορές. Υπό το παρόν οικονομικό ε, κλίμα. Είναι σημαντικό ο κόσμος να έχει εμπιστοσύνη στις ε, ε, αγορές και θα πρέπει να έχουμε αρκετά μέσα, αποτελεσματικά μέσα για να αποτρέψουμε τις εγκληματικές ενέργειες. Έχουμε δει τα τελευταία χρόνια τις καταστροφικές επιπτώσεις ατομικών πράξεων στις οικονομικές αγορές όπως είναι οι ενέργειες της στιγμή που κατέχονται εμπιστευτικές πληροφορίες ή οι, οι παρόμοιες ενέργειες. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι οι ποινικέ κυρώσεις θα είναι απαραίτητο μέτρο για να καταπολεμήσουμε τα βασικότερα αδικήματα στις οικονομικές αγορές και είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής μας για την χειραγώγηση της αγοράς. Προτείνουμε λοιπόν ένα ε, Εξετάσαμε μάλλον ε, το καθεστώς στα διάφορα και βλέπουμε μια μεικτή εικόνα. Μεγάλος αριθμός ε, κρατών μελών έχουν ποινικέ κυρώσεις ε, στο εθνικό δίκαιο για κάποιες εγκληματικές πράξεις που συνδέονται με την αγορά. Αλλά δεν τιμωρούν όλα την κατοχή εμπιστευτικών πληροφοριών και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. Επίσης, Υπάρχουν σημαντικέ αποκλήσει ε, στον ποινικό κανόνα των διαφόρων κρατών μελών. Η κατάσταση λοιπόν διαφέρει ε, από χώρα σε χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθότι η ε, χειραγώγηση τη αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί διασυνοριακά. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να υπονομεύσει και κάποιε πτυχέ τη εσωτερική αγορά. Η ανάλυση μα λοιπόν δείχνει ότι τα πιο προφανή προβλήματα είναι ότι δεν έχουν ποινικοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη τη χειραγώγηση τη αγορά και τις και ότι οι ορισμοί διαφέρουν από κράτο μέλο σε κράτο μέλο, ε, κάτι που οδηγεί σε κατακαιρματισμό. Έχουμε λοιπόν προτάσει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά ε, με την ε, Συμφωνία Κοινών Ορισμών για τη χειραγώγηση της αγοράς και τις συναλλαγές ατόμων που κατέχουν πιστευτικές πληροφορίες. Έχουμε λοιπόν αναλογικά και αποτρεπτικά μέτρα. Έχουμε εφαρμόσει πολύ αυστηρά την αρχή της αναλογικότητας και γι' αυτό δεν προτείνουμε τίποτα παραπάνω από ό,τι θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουμε την ε, αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής μας. Πιστεύουμε ότι οι ελάχιστες κυρώσεις ε, θα έχουν ισχυρό αποτρεπτικό χαρακτήρα και θα ε, βοηθήσουν να διασφαλιστεί η ακαιρεότητα των οικονομικών αγορών στην Ευρώπη και ότι έτσι θα έχουμε και αποτελεσματική εποπτεία τη εφαρμογή τη πολιτική μας. Ε, λέμε ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες ε, ε, αποτρεπτικές και έχουμε εξετάσει προβλέψει έκθεση προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μετά από τέσσερα χρόνια εφαρμογής της οδηγίας. Ε, με στόχο να ε, θεσπιστούν ελάχιστοι κανόνες όσον αφορά ε, τον τύπο και το επίπεδο των ποινικών κυρώσεων. Πιστεύουμε ότι αυτή η προσέγγιση είναι κατάλληλη για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων για την χειραγωγήση των αγορών. Ε, είμαι βέβαιη ότι θα αναγνωρίσετε ε, διατάξεις που προέρχονται από προηγούμενες ε, προτάσεις όσον αφορά την ευθύνη νομικών προσώπων, τα στοιχήματα και άλλες πράξεις. Πάντως γενικά στην αξιολόγησή μας πιστεύουμε ότι με τις ποινικέ κυρώσεις στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα αυτή τη στιγμή για να αποτρέψουμε ε, πιθανούς εγκληματίες ε, και ε, δείχνουμε ότι είμαστε σοβαροί όσον αφορά την καταπολέμηση της χειραγώγησης της αγοράς. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σήμερα στους πολίτες μας ώστε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη στις αγορές. Είναι λοιπόν πρώτη φορά που έχουμε μια τέτοια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 83.2 ε, πρόκειται δηλαδή για μέσο του ποινικού δικαίου και ε, προσβλέπουμε στην ε, καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα την Επιτροπή ΛΙΝΤΕ για να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Η κυρία Μπόκετ που είναι η συγγετριά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ βάθους καρδίας για την παρουσίαση που μας έκανε. Συμφωνώ απόλυτα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν όταν λέει ότι θα πρέπει να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη στις, προς για να το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να αποφύγουμε χειραγώγηση των αγορών και να έχουμε μια κοινοτική στάση. Διότι πρόκειται για διασυνοριακές ε, δραστηριότητες, ε, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης ε, απέναντι στους καταναλωτές, διότι όποιος διαπράττει αυτά τα εγκλήματα δεν θα πρέπει να μπορεί να ξεφεύγει ατιμόρυτος. Υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα καθαρά. Ε, να θέσω λοιπόν σε τούτου κάποια ερωτήματα. Το ζήτημα της ε, αναθεώρησης ε, η Κομισιόν είπε πως ε, θα πρέπει να επανεξεταστεί μετά από τέσσερα χρόνια. Τέσσερα χρόνια ίσως να είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί επιλέξατε τέσσερα χρόνια Κομισιόν Γιατί επιλέξατε λοιπόν αυτή την χρονική διάρκεια τη τετραετία. τώρα, στο 3, άρθρο 3-4. Στο άρθρο 3 λοιπόν, πώς ε, μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα πράγματα είναι σαφή και απόλυτα κατανοητά. Τώρα στο άρθρο 5 αναφέρεται πως ε, αυτή η χειραγώγηση της αγοράς ε, λοιπόν και τι εννοείται σε αυτό το πλαίσιο πρόσωπα που κατέχουν εμπιστευτικές ε, πληροφορίες Και κάτι ακόμα. Οι κυρώσεις, κυρώσεις. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι αποτελεσματικές, αποτρεπτικές. Υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα, αλλά θα σας τα θέσω σε άλλη περίσταση. Ακούσαμε λοιπόν κάποιες ε, ερωτήσεις. Ε, η Κομισιόν μπορεί να απαντήσει παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι ρωτήσεις ε, δείχνουν ότι γνωρίζετε το ζήτημα. Τώρα τα, η τετραετία. Αυτό οφείλεται στο ότι τα κράτη-μέλη έχουν 24 χρόνια για την μεταφορά του στο ιστορικό δίκαιο. Λοιπόν, 24 μήνες ε, μέχρι να μεταφερθεί στην ε, εθνική νομοθεσία και μετά χρειάζεται να εξετάσουμε τα αποτελέσματα. Πρέπει να αναλύσουμε λοιπόν πώς ε, η εθνική νομοθεσία λειτουργεί μετά από την ε, μεταφορά αυτής της οδηγίας και να δούμε κατά πόσον οι αποτρεπτικές ε, και αποτελεσματικές κυρώσεις έχουν πετύχει το στόχο τους. Επίσης, δεδομένου ότι αυτό είναι ένα νέο πεδίο για το ποινικό δίκαιο, εάν ε, θελήσουμε να ακολουθήσουμε τον δρόμο των κυράσεων, θα πρέπει να το μελετήσουμε το ζήτημα πολύ προσεκτικά. Όπως γνωρίζετε από το παρελθόν, μια συγκριτική μελέτη θα πρέπει να γίνει στα κράτη-μέλη για να δούμε τι είδους κυρώσεις έχουν και εφαρμόζουν και τι κυρώσεις συνήθως που χρειάζονται για να πετύχουμε την επιθυμητή ε, λειτουργία των κυρώσεων αυτών. Τώρα για το incitement που αναφέρατε είναι κάτι το οποίο ε, μπει στο πλαίσιο του ποινική διαδικασία. Ε, είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν στους ορισμούς ε, των σημείων 3 και 4 για να χρησιμοποιήσουμε μια ποινική ορολογία και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το ζήτημα της, ε, του επηρεασμού των αγορών και της χειαγώγης αγοράς είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο πλαίσιο του Συμβουλίου αυτή την περίοδο και θα φροντίσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ε, αλλαγές αλλά είναι κάπως νωρίς ακόμα. Θα πρέπει λοιπόν ο Εθνικός Δικαστής να κρίνει και να ορίσει αυτό το incitement ε, αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Τώρα, οι ρυθμίσεις ε, που αφορούν στη χειραγώγηση της αγοράς ε, προβλέπουν κυρώσεις που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο. μην ξεχνάμε ότι στα τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετική νομοθεσία, υπάρχει διαφορετικό ποινικό δίκαιο, αλλά παντού ισχύει το nebis in idem σε όλα τα δικαιάκα συστήματα. Και αυτό για να αποφύγουμε ε, διπλές κυρώσεις. Τώρα, για τον προσδιορισμό κατά πόσον εμπίπτει ε, σε ποινικό αδίκημα ή όχι, υπάρχει ένα κατόφλι μετά από το οποίο η πράξη θεωρείται ως ποινικό αδίκημα, αλλά εμπεστώσει και εδώ ο εθνικό Δικαστής είναι αυτός ο οποίος ε, θα το κρίνει. Ευχαριστώ. Thank you. about Θέλετε κυρία Σιγητρία, να θέσετε ερωτήματα. Όχι. Όχι άλλη λοιπόν ανάκριση. Ωραία. Εντάξει. Κατά την παράσταση εξέταση. Ολοκληρώνουμε λοιπόν με το θέμα αυτό. Το θέμα είναι σίγουρα σημαντικό. Και εγώ έτσι σκέφτομαι ότι πρέπει να το δούμε και από την πλευρά της διαδικασίας. Θα πρέπει να τονίσουμε αυτό το ζήτημα και άλλη μια επιτροπή ασχολείται. Ξεκινάμε όμως, ακούσαμε την παρουσίαση της Επιτροπής και είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψε με την εισηγήτρια που μόλις ορίστηκε. Αλλά δεν ε, θα προχωρήσουμε άλλο σήμερα, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Συνεδριάσαμε 15 ώρες στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ σήμερα και χθε. Εντάξει, ποτέ δεν είναι αρκετά, αλλά τουλάχιστον για σήμερα είναι αρκετά. Γεια σας.